Witam Państwa z Αγαπητοί συνάδελφοι, καλημέρα σας. Έχουμε ήδη καθυστερήσει πέντε λεπτά. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν τη συνεδρίασή μας. Να σας πω καταρχάς ότι εγώ έφτασα πριν από 20 λεπτά σε αυτή την αίθουσα. Περίμενα λοιπόν 20 λεπτά και ακόμα υπάρχουν μέλη της Επιτροπής μας που δεν έχουν φτάσει. Θα πρέπει λοιπόν να καλύψουμε την καθυστέρηση αυτή και ελπίζω θα το κάνουμε αυτό ψηφίζοντας γρήγορα και αποτελεσματικά. Σας καλωσορίζω λοιπόν. Και θα ήθελα καταρχάς να σας ενημερώσω για το τι θα κάνουμε σήμερα. Καταρχάς, όσον αφορά το σημείο 16 της ημερήσιας διάταξης που έχει να κάνει με τον προπολογισμό, θα αναβληθεί στην επόμενη συνεδρίαση που θα έχουμε τον Ιούλιο. Αιτιολογούν διάφοροι λόγοι την αλλαγή αυτή. Υπάρχουν πολλοί βουλευτές οι οποίοι θα πάνε στο Μιλάνο σήμερα που πρέπει να αποχωρήσουν. Λοιπόν, έχει εγκριθεί, φαντάζομαι, η αλλαγή αυτή, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Μπορούμε να περάσουμε λοιπόν ευθύ αμέσω στις ε, ψηφοφορίες. να ξεκινήσουμε την έκθεση για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης προς ελέγχους βάση απόδοση στην κοινή αγροτική πολιτική. Ο κύριος και είναι ο εισηγητής. Αρμόδια καθήλυν επιτροπή είναι η Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού. Θα μπορούσαμε να δώσουμε καταρχάς το λόγο στον κύριο Σαρβαμά, ο οποίος γνωρίζει πολύ καλύτερα το ζήτημα αυτό από ότι εγώ. Είναι όμως παρόν στην αίθουσα ο κύριος Σαρβαμά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ο, ο συνάδελφο Άρβαμα δεν είναι εδώ, νομίζω. Κάνουμε την γνωμοδότηση από την Επιτροπή Προπολογισμού. Έχουμε πάνω από 120 τροπολογίες, αλλά δεν υπάρχει πρόβλημα, θεωρώ. Μπορούμε να περάσουμε πάρα αυτά στην ψηφοφορία. Πολύ ωραία. Λοιπόν, αν δεν υπάρχουν άλλε παρατηρήσει ξεκινάμε την ψηφοφορία. Συμβαστική τροπολογία Α, με ηλεκτρονική ψηφοφορία παρακαλώ. Ο κύριος Νταντών ξέχασε την κάρτα του, το καταγράφουμε. Συμβαστική τροπολογία Α, άρχεται ψηφοφορία. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά παρακαλώ. Πέρας. Εγκρίνεται. Και πρέπει βέβαια να προσθέσουμε εδώ πέρα και την ψήφο του κύριου Νταντά. Περνάμε στην τροπολογία 35. με τα σχηρώσει υπέρ παρακαλώ κατά απορρίπτεται 36 υπέρ εγκρίνεται Περνάμε στη βασική τροπολογία Β, άρτη ψηφοφορία, ψηφίζουμε ηλεκτρονικά παρακαλώ. Πέρας. Εγκρίνεται ομόφωνα. Και βέβαια προφανώς καταγράφουμε και την ψήφο του κύριου Νταντά. Περνάμε τώρα στην 43 ε, του κύριου Καπούτο, υπέρ παρακαλώ. Κατά. Απορρίπτεται. 44 υπέρ παρακαλώ. Κατά. Απορρίπτεται. 45 υπέρ. Εγκρίνεται. 46 υπέρ. Εγκρίνεται. 47 υπέρ παρακαλώ. Εγκρίνεται. Τροπολογία 48 υπέρ. Εγκρίνεται. Τροπολογία 49 υπέρ παρακαλώ κατά, απορρίπτεται. Τροπολογία 50 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Θέλετε να επαληθεύσουμε αυτή την τροπολογία, όχι. Άρα περνάμε στη συμβαστική τροπολογία Γ σε άρτη ψηφοφορία. Πέρας. Υπεράριθμοι από το ECR παρακαλώ. Ψηφίζει ένας επιπλέον. Εγκρίνεται η συμβαστική τροπολογία C. Περνάμε στην τροπολογία 59 υπέρ κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 60 υπέρ κατά Απορρίπτεται. Τροπολογία 61 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 62 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 63 υπέρ παρακαλώ. Κα... Εγκρίνεται. Τροπολογία 64 υπέρ. Εγκρίνεται. 65 υπέρ. Κατά. Νομίζω ότι έχει απορριφθεί, αλλά θα το παληθεύσουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία για τροπολογία 65. Πέρας. Όντως απορρίπτεται. Τροπολογία 66 υπέρ. Εγκρίνεται. Τροπολογία 67 υπέρ εγκρίνεται. Τροπολογία 68 υπέρ κατά απορρίπτεται. Τροπολογία 60 μαλε 70 υπέρ εγκρίνεται. Τροπολογία 71 υπέρ κατά Νομίζω ότι έχει εγκριθεί, αλλά θα το επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά, σας παρακαλώ. Ψηφίσουμε ηλεκτρονικά για την τροπολογία 71, πέρας. Απορρίπτεται. Με μικρή διαφορά βέβαια. 72 υπέρ. Κατά. Θα επαληθεύσουμε και την τροπολογία 72 ηλεκτρονικά, άρτη ψηφοφορία. Πέρας. Πάλι από τους σοσιαλιστές υπεράριθμοι. Πέρας. Λοιπόν, επαναλαμβάνουμε σα παρακαλώ πολύ την ηλεκτρονική ψηφοφορία για την τροπολογία 72. Άρθη ψηφοφορία. Πέρα. Εγκρίνεται. Κύριε για μην αποσπάτε τους συναδέλφους σας. 73 υπέρ. Εγκρίνεται. Τροπολογία 74 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 75 υπέρ παρακαλώ. Κατά. Απορρίπτεται. 76 υπέρ. Εγκρίνεται. Περνάμε σε συμβαστική τροπολογία D. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά άρτη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Και προφανώς για άλλη μια φορά καταγράφουμε και την ψήφο του κύριου Νταντά. 87 από την τροπολογία 87 ως 91 on block υπέρ κατά απορρίπτονται. Αν δεν θέλετε την ομαδική αυτή ψηφοφορία, λοιπόν, ξεχωριστά, 87 παρακαλώ υπέρ, κατά, απορρίπτεται, τροπολογία 88 υπέρ, κατά, απορρίπτεται, Τροπολογία 89 υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονική επαλήθευση για τροπολογία 89 άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 90. Υπέρ κατά. Ηλεκτρονική επαλήθευση για την τροπολογία 90 άρτη ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 91. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία ε ή άρτη ψηφοφορία. Ψηφίσουμε ηλεκτρονικά παρακαλώ. Πέρας. Εγκρίνεται. Περνάμε στην τροπολογία 95. Υπέρ παρακαλώ. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία F, άρτη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 103. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 104. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 105 υπέρ ηλεκτρονική επαλήθευση για την τροπολογία 104, άρτη ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται 105 υπέρ. Εγκρίνεται. 106 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 107 υπέρ. Εγκρίνεται. Τροπολογία 108 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 109 υπέρ. Εγκρίνεται. Μπορούμε να ψηφίσουμε ομπλόκ block όλες τις τροπολογίες κυρίας Σκοτ κάτω ή θέλετε να τις ψηφίσουμε τελικά χωριστά. Από την 110 ως την 120, ξεχωριστά σε κάθε περίπτωση την 121. Από την 110 έως την 120 on block. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Απορρίπτονται. Τροπολογία 121 υπέρ. Εγκρίνεται. Τροπολογία υπαριθμών 1 υπέρ. Εγκρίνεται. Τροπολογία 2 υπέρ. Εγκρίνεται. Τροπολογία 3 υπέρ. Εγκρίνεται. 4 υπέρ. Εγκρίνεται. Τροπολογία 5 υπέρ. Εγκρίνεται. Τροπολογία 6. Υπέρ. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία G. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 12. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 13 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 14 υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονική επαλήθευση για τροπολογία 14 άρτη ψωφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Με μία ψήφο διαφορά βλέπετε ότι σε κάθε περίπτωση αν υπάρχει οποιαδήποτε αμφιβολία φροντίζω να κάνω ηλεκτρονική επαλήθευση. Ήσασταν και εσείς κατά ούτως άλλως το αποτέλεσμα δεν αλλάζει. Τροπολογία 15. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 16. Υπέρ εγκρίνεται. Τροπολογία 17 υπέρ κατά απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία H μάλλον όχι. Θα επαληθεύσουμε πρώτα την τροπολογία 17. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά άρχιδη ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία H Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Άρχιδη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίθηκε ομόφωνα. Τροπολογία 21 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Μπορούμε να ψηφίσουμε on μπλοκ ε, της... Ε, μάλλον όχι την 22 πρώτα, υπέρ παρακαλώ, υπέρ της τροπολογίας 22 εγκρίνεται. Μπορούμε να ψηφίσουμε από κοινού τις υπόλοιπες τροπολογίες. Όχι, μάλλον λοιπόν 23 υπέρ, κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 24 υπέρ, κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 25 υπέρ, κατά Θεωρήσω τμήμα τη αίθουσα δεν σηκώνετε τα χέρια σα, επομένω επαληθεύουμε ηλεκτρονικά για την τροπολογία 25. Άρτη ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Με μία μικρή διαφορά ψήφων. Περνάμε στην τροπολογία 26. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Απορρίπτεται. Περνάμε τώρα στην ψηφοφορία για το σύνολο του κειμένου όπως τροποποιήθηκε. Ψηφίσουμε ηλεκτρονικά άρχιδη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ για τη βοήθειά σας. Τώρα θα περάσουμε στην έκθεση της κυρίας Πόλσεν. Χθες η Ευρωβουλευτής μας παρουσίασε την έκθεσή της. Την έχουμε ήδη ευχαριστήσει και συγχαρεί. Θέλετε να πάρετε το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Από ό,τι φαίνεται δεν έχετε κάτι άλλο να προσθέσετε. Ας περάσουμε λοιπόν στην ψηφοφορία. Θα ψηφίσουμε λοιπόν το αποτέλεσμα του τριμερούς διαλόγου. Με ονομαστική κλίση άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Θα ήθελε κάποιος να πάρει το λόγο για αυτό το θέμα. Όχι, ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εντάξει, μπορούμε να περάσουμε στο σημείο 11 λοιπόν. παρουσίαση της μελέτης για την έκταση του φαινομένου της υφαρπαγής γεωργικών γεών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ξεκινήσουμε με την ε, παρουσίαση του ζητήματος αυτού για την έκταση δηλαδή αυτού του φαινομένου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ok. Myślę, że już wystarczy tej Εντάξει, αφήσαμε και ένα λεπτό για να φύγουν όσοι ήθελα, να περάσουμε λοιπόν στο θέμα μας. Η μελέτη αυτή λοιπόν αφορά την έκταση του φαινομένου της εφαρπαγής γεωργικών γεών. Πολλά στοιχεία δείχνουν ότι η εφαρπαγή γεωργικών γεών είναι ένα ε, φαινόμενο που λαμβάνουμε όλο ένα και μεγαλύτερε διαστάσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή η μελέτη διερευνά τι αιτίε αυτή τη πρακτική και αναλύει και την επιρροή ε, τη εφαρπαγή ε, γεών στην επιστηστική ασφάλεια και ανεξαρτησία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον αντίκτυπο στην απασχόληση ε, στις γεωργικές περιοχές και για το περιβάλλον βεβαίως. Η μελέτη αυτή αναφέρει ότι η χαρπαγή γεών, ιδίως ε, όταν αυτό το φαινόμενο συνδέεται με άλλα κρίσιμα ζητήματα, ε, γεωργικά και το καθεξής, χρήζουν Μία ε, ορθής μεταρρύθμισης του τομέα αυτού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα να συγχαρώ και να καλωσορίσω τους ε, συγγραφεί αυτής της μελέτης, την κυρία Σίλβια Κέι και τον κύριο Τζόναθαν Πέιτς. Ως ήθιστε, πριν από τη συζήτηση θα δώσουμε το λόγο στους εμπειρογνώμονές μας και στη συνέχεια θα ακούσουμε τα μέλη. Εσείς μπορείτε να διαλέξετε ποιος θα μιλήσει πρώτος. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Πρώτα απ' όλα θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την Κοινοβουλευτική Επιτροπή ε, Γεωργικών Υποθέσεων ε, και Ανάπτυξης Υπαίθρου που αναθέσατε αυτή τη μελέτη στο Ινστιτούτο μας για ένα τόσο ενδιαφέρον και ανησυχητικό ζήτημα. Ονομάζομαι Σιλβία είμαι ερευνήτρια στο TNI, το Transnational Institute, που είναι ένα διεθνές αισθητούτο που εξετάζει ε, μία σειρά ε, παγκοσμίων πολιτικών, επιστημική ασφάλεια, ε, διαχείριση φυσικών πόρων και ούτω καθεξής. Να δώσω το λόγο και στον συνάδελφο για να σας συστηθεί, εφόσον από κοινού παρουσιάζουμε αυτή τη μελέτη. Καλημέρα, Τζοναθάν Πέτσο ονομάζομαι και εγώ είμαι ερευνητή στο TNI και θα παρουσιάσω κάποια ζητήματα που αφορούν τις ε, γεωργικές γέες στην Ευρώπη. Ένα από τα κύρια ζητήματα που θα σας παρουσιάσουμε σήμερα είναι ότι κατά τη γνώμη μας η υφαρπαγή γεωργικών γεών, παρότι από μόνο τους ως φαινόμενο είναι εξαιρετικά ανησυχητικό, αντιμετωπίζει και βαθύτερα ζητήματα όπω είναι η διανομή στην πρόσβαση και η χρήση και έλεγχο των γεωργικών νεών. Και έτσι αυτό έχει μια νέα προσέγγιση, απαιτεί μάλλον μια νέα προσέγγιση στην χρήση γεωργικών νεών ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να σα παρουσιάσω πρώτα τη δομή. Πρώτον θέλουμε να ε, παρουσιάσουμε κάποια προκαταρκτικά πορίσματα τη μελέτη, ό,τι αφορά την κλίμακα, το πεδίο εφαρμογή και το χαρακτήρα της υφαρπαγής γεών στην Ευρώπη. Μετά θα αναφέρουμε κάποιους ε, βασικούς ε, κινητήρους μοχλούς που ε, δημιουργούν ένα ευνοϊκό περιβάλλον, αν θέλετε, για την υφαρπαγή γεών στην Ευρώπη. Μετά θέλουμε να συνδέσουμε την υφαρπαγή γεών με άλλα κρίσιμα και φλέγοντα ζητήματα χρήση γης στην Ευρώπη, όπως είναι η συγκέντρωση της γεωργικής γης. Και τέλος, θα παρουσιάσουμε και κάποιες ε, συστάσεις πολιτικής και εναλλακτικέ λύσεις ε, για την αντιμετώπιση του φαινομένου. Για τα αρχικά μας λοιπόν ε, πορίσματα, πριν σας τα παρουσιάσω, κάποια σύντομα μεθοδολογικά σχόλια. Δεν θα επισέλθω σε λεπτομέρειε γιατί φαντάζομαι και σας τα γνωρίζετε αλλά για να σας ε, αναφέρω ορισμένες προκλήσεις με τις οποίες ήρθαμε αντιμέτωποι. Σίγουρα ξέρετε ότι ε, οι απόψεις δείστε σε ό,τι αφορά τον ορισμό της εφαρπαγής. Αυτό που για κάποιον είναι μια ε, παραγωγική επένδυση, για κάποιον άλλον είναι εφαρπαγή γεών. Μετά υπάρχει έλλειψη διαφάνειας σε ό,τι φορά και την συλλογή δεδομένων και πολύ συχνά επικεντρωνόμαστε στο γεγονός ότι ε, είναι οι ξένοι επενδυτέ που φταίνε ε, για την φαρπαγή γεών, όμω, αυτό δείχνουν, οι μελέτες δείχνουν ότι και οι εγχώροι ε, είναι αυτοί που προβαίνουν στην φαρπαγή. Και επίση υπάρχει υπόθεση ότι η Ευρώπη κάπως δεν την αφορά την Ευρώπη αυτό το ζήτημα. Δηλαδή ότι λιγότερη έμφαση έχει δοθεί στην υφαρπαγή γεωργικών γεών στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι τώρα. Τουλάχιστον εμεί με αυτή τη μελέτη έχουμε διορθώσει αυτή την υπόθεση. Υπάρχει φαρπαγή γεωρικών γεών στην Ευρώπη και είναι κάτι το οποίο επηρεάζει και το ευρωπαϊκό κεφάλαιο, τι ευρωπαϊκέ γέ και ε, τον ευρωπαϊκό πληθυσμό. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτή τη μελέτη εμεί εκπονήσαμε και έναν ορισμό από ευρωπαϊκή σκοπιά, θεωρούμε ότι αυτό είναι σημαντικό. Η χαρπαγή γεών λοιπόν στην Ευρώπη αφορά ορισμένες ε, συμφωνίες που είναι εκτός ε, ευρωπαϊκής κλίμακας και αναλογίας και έτσι ε, δημιουργούμε δομές με χιλιάδες εκτάρια γης. Δεύτερον, έχουμε τον έλεγχο της λήψης αποφάσεων σε μία χώρα, όπως είναι για παράδειγμα φυσική πόρη, ποιος θα χρησιμοποιεί τις για ποιον σκοπό και για πόσο χρονικό διάστημα υπονοούν και μία υπερβολική οικονομική ισχύ και έτσι οδηγείται στη συγκέντρωση. Υπάρχουν και κάποια εξτρά λοιπόν κίνητρα, ακόμα και με δικού όρου που παρέχονται από το κράτο, με καλέ ε, διασυνδέσει πολιτικέ, στήριξη κυβερνήσεων και διάφορες μορφές παράκαμψη του νόμου. Και τέλος, όπως σημειώνει και η ΕΟΚΕ, η φαρπαγή γεών δείχνουν ότι υπάρχει μία σαφής ρήξη ε, με, με το σύνηθες ευρωπαϊκό μοντέλο της οικογενειακής ε, καλλιέργειας ε, και τον στόχο της διαφοροποιημένης γεωργίας. Να σας παρουσιάσω λοιπόν κάποια πρώτα βασικά πορίσματα σε ό,τι αφορά την κλίμακα. Εξετάσαμε πολλά σύνολα δεδομένων σε διεθνές επίπεδο για τις ε, μεγάλες κλίμακες ε, γεωργικές ε, συμφωνίες ε, παγκοσμίω, όμως κάποια στοιχεία έλειπαν σε ό,τι φορά την Ευρωπαϊκή Έχουμε το Land Matrix Database που από το Μάρτιο του 2015 έχει καταγράψει τέτοιες μεγάλες κλίμακες συμφωνίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση με σύνολο 166.359 εκτάρια. Όμως εμείς θεωρούμε ότι ε, υποτιμάται η πραγματική κλίμακα της υφαρπαγής γεωργικών γεών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε δει και διάφορα συμπληρωματικά στοιχεία. Η Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινωνική Επιτροπή έχει συλλέξει τέτοια στοιχεία, αλλά και διάφορες, 13 ε, μάλλον τον αριθμό case studies, ε, που εξέτασε το TNI από τη Συμμαχία Κάτω τα Χέρια από τη Γη και δείχνουν ότι πέρα ε, των ε, ε, επισήμων δεδομένων υπάρχουν πολλές άλλες περιπτώσεις φαρπαγιδιών, όπως υπάρχουν κάποιες τα λεγόμενα pocket contracts στην Ουγγαρία ή εικονικοί αγοραστές στην Πολωνία. Είναι ένα φαινόμενο που υπάρχει τις τελευταίες δύο δεκαετίες. Οι εικονικοί αγοραστές ε, στην ε, Πολωνία, dummy buyers, είναι Πολωνοί υπήκοοι, μικροί καλλιεργητές συνήθως, που έχουν, πληρούν τα βασικά κριτήρια για να έχουν μια, μια προσωρινή κατοχή γης και ε, αφήνουν μια εταιρεία να αγοράσει το, τη γη, παρότι υπάρχει απαγόρευση με βάση το πολωνικό δίκαιο. 200.000 εκτάρια γης έχουν αγοράσει ξένοι επενδυτές στην Δυτική Πομερανία με αυτούς τους εικονικούς αγοραστές. Θέλω να πω ότι παρότι μπορεί να φαίνεται ότι η φαρπαγή γεών στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αμεληταία, η πραγματική κλίμακα δεν μπορεί να φανεί ξεκάθαρα από αυτά ε, τις βάσεις δεδομένων. Και υπάρχουν σημαντικά στοιχεία που δείχνουν ότι το φαινόμενο είναι πολύ ευρύτερο. Δεύτερον τώρα, για το πεδίο εφαρμογή. Βλέπουμε ότι η εφαρμογή γεών ε, παρουσιάζει ανισομετρίες ε, στην Ευρώπη. Συνήθως, αλλά όχι αποκλειστικά, συγκεντρώνονται στην Ανατολική Ευρώπη. Έχουμε πει τέτοιε περιστάσεις, ιδίω περιστάσεις Ρουμανία, Βουλγαρία, Ουγγαρία και σε έναν βαθμό και στην Πολωνία. Σε ό,τι αφορά το χαρακτήρα αυτής της ευρωπαϊκής γης βλέπουμε ότι πολλοί ε, περιλαμβάνουν νέα σύνολα παραγόντων ή φορέων, είτε από τον χρηματοπιστωτικό τομέα, τράπεζες, ακόμα και ε, δεξιωτικά ταμεία και το καθεξής, αλλά και οι λεγόμενοι land brokers, πολλές φορές είναι μια εσωτερική ελίτ ε, με συγκεκριμένα συμφέροντα για τη γη. Και όπως ανέφερα και προηγουμένως, πολλές από τις ε, περιπτώσεις εφαρπαγές αφορούσαν ε, γεές τεράστιας κλίμακας. Για παράδειγμα, υπάρχει μία έκταση 65.000 νεκταρίων ε, γης. Κάποιοι θεωρούν ότι η καλύτερη περιγραφή είναι ένα περιορισμένο αλλά και ανησυχητικό φαινόμενο που ε, επεκτείνεται σταδιακά. Είναι ας πούμε ίσονο σημασία σε σχέση με την Αφρική, όμως αυξάνεται γιατί υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν ότι άμα το αφήσουμε ανεξέλεγκτο θα μπορούσε να επιταχυνθεί και να επεκταθεί γρήγορα. Για παράδειγμα, στη Σερβία, στην Ουκρανία θα μπορούσαμε να το εξετάσουμε περαιτέρω ε, ή αν αυτό συνδεθεί περαιτέρω με άλλε συνεργασ... με άλλες διεργασίες συγκέντρωσης Γιατί υπάρχει και η γενική τάση συγκέντρωση τη γη και είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να απασχολήσει και ε, τον τομέα τη πολιτική. Euh, merci Sylvia. Donc nous allons maintenant aborder la question du cadre réglementaire. Τώρα θα περάσουμε στο κανονιστικό πλαίσιο και ιδίως σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, για τις ε, γεωργικές γέες. Αναφερόμαστε σε τέσσερι πολιτικέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση που μπορεί να έχουν επίπτωση στην έγκυο ιδιοκτησία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε την κοινή γεωργική πολιτική, τον κανονισμό τη εσωτερική αγορά, την περιβαλλοντική πολιτική, καθώ επίση και την πολιτική τη χωροταξία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα αναφερθώ τώρα στο καθεστώ που υπάρχει όσον αφορά την εσωτερική αγορά και την κοινή γεωργική πολιτική. Όσον αφορά την κοινή γεωργική πολιτική, ποια είναι η σχέση με τι γεωργικέ γέε Πολλέ μελέτε τα τελευταία χρόνια κατέδειξαν την επίδραση τη κοινή γεωργική πολιτική στην διοκτησία γης, διαφορετικές επιπτώσει αυτέ και ιδιαίτερα σοβαρέ. Πολύ συχνά μα λένε ότι ε, δεν επηρεάζει ουσιαστικά η πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση στην διοκτησία γη. στην πράξη όμω έχουμε τα πράγματα εντελώ διαφορετικά. Καταρχά βλέπουμε ότι έχουμε άμεσε ενισχύσει που δίνονται προ τι γεωργικέ εκτάσει. Ξέρετε ότι είναι κάτι το οποίο έχουμε κληρονομήσει από την προηγούμενη ΚΑΠΑ, ισχύει και στην υφιστάμενη και επιπτώσεις παραμένουν. Βλέπουμε ότι επηρεάζει το οικονομικό μέγεθος της γεωρικής εκμετάλλευσης, τον τύπο της παραγωγής, την ίδια την έκταση της γεωρικής εκμετάλλευσης, καθώς επίσης και τον τύπο της σύμβασης μπορεί να υπάρχει ανάμεσα στον ιδιοκτήτη και την ίδια τη γη. Οπότε μιλάμε για μίσθωση, για ιδιοκτησία γης. Βλέπετε εδώ πέρα στη γραφική παράσταση που έχουμε στην οθόνη το τμήμα εκείνο της κοινή γεωργικής πολιτικής και το πώς επηρεάζει διάφορες χώρες. Βλέπουμε ότι για παράδειγμα στη Ρουμανία τα πράγματα είναι αρκετά δραματικά. 1% των γεωκτημόνων στη χώρα αυτή εποφελούνται από το 50 περίπου των άμεσων ισχύσεων της κοινή γεωργικής πολιτικής. Λοιπόν, ποια είναι τα αποτελέσματα της ε, τάσης αυτής. Πρώτον, όσο μεγαλύτερη είναι η γεωργική εκμετάλλευση, τόσες περισσότερες ενισχύσεις λαμβάνει, επομένω θα αυξάνεται όλο και περισσότερο. Οι μεγαλύτερε γεωργικέ εκμεταλλεύσει λοιπόν βρίσκονται σε θέση υπεροχή όσον αφορά την παγκόσμια αγορά. Επίση, έχουμε μία μείωση των μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην Ευρώπη. Στη γραφική παράσταση βλέπετε ότι μεταξύ του 2005 και του 2006 τα αγροκτήματα τα οποία είναι κάτω από τα 5 εκτάρια έχουν χάσει ένα 3% των εισοδημάτων τους, ενώ οι μεγάλες ζωρικές εκμεταλλεύσεις όλο και αυξάνονται. Ξέρετε επίσης ότι υπάρχει και ένα κατόφλι 5.000 ευρώ όσον αφορά τα έσοδα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων προκειμένου να λάβει κανεί άμεσε ενισχύσει. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι οι άμεσε ενισχύσει τελικά πηγαίνουν στι μεσαίε και μεγάλε γεωργικέ εκμεταλλεύσει, ενώ διόλου δεν αποφελούνται οι μικρέ γεωργικέ εκμεταλλεύσει. Βλέπετε επίση στα πλαίσια της κοινή γεωργικής πολιτικής ότι υπάρχουν διάφορες αρνητικές επιπτώσεις. Βλέπουμε ότι πολύ συχνά οι ενισχύσει πηγαίνουν μόνο σε εξειδικευμένες γεωργικές εκμεταλλεύσεις με εξειδικευμένες καλλιέργειες, δεν προσφέρουν πολλές θέσει απασχόληση και πειράζουν επίση πολύ αρνητικά και το περιβάλλον. Καταλαβαίνετε ότι κάτι τέτοιο είναι ιδιαίτερα αρνητικό στα πλαίσια της ε, κλιματικής, της κατάστασης κλιματικής αλλαγής την οποία αντιμετωπίζουμε. Νομίζω ότι θα πρέπει να είχαμε μια κοινή γεωργική πολιτική η οποία να ωφελεί περισσότερο τις μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις, πραγματικά να δημιουργεί θέσεις απασχόλησης ε, στην Ήπεθρο και να οδηγεί στην παραγωγή προϊόντων τη προστιθέμενης αξίας, πραγματικά θα έχουν ευνοϊκή επιρροή στους τοπικούς πληθυσμούς και στις τοπικές περιφέρειες. Ας περάσουμε τώρα στην ε, δεύτερη πολιτική που πειράζει την έγκυο ιδιοκτησία, την εσωτερική αγορά. Η εσωτερική αγορά δημιουργεί το σημαντικότερο πλαίσιο ιδιοκτησίας γης. Η ε, γη θεωρείται ως ε, ακίνητη περιουσία, ως περιουσιακό στοιχείο, αυτά άλλωστε έχει πει και το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης απόφασή του. Επομένως μπορεί οποιαδήποτε γη να αγοραστεί από οποιονδήποτε αγοραστεί επενδυτή εντός ή εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποια είναι η βασική αρχή της εσωτερικής αγοράς, το να καταρρύψει οποιοδήποτε εμπόδιο υπάρχει στις τέσσερις βασικές ελευθερίες. Ελεύθερη δηλαδή διακίνηση κεφαλαίων, ανθρώπων, προϊόντων και υπηρεσιών. Κατά αυτόν τον τρόπο λοιπόν γίνεται ένα απλό προϊόν το οποίο μπορεί να πουληθεί, να αγοραστεί. Αυτό είναι πλέον, αυτή είναι η μοίρα που επιφυλάσσεται για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια της ιστορικής αγοράς. Δυστυχώς όμως και εδώ πέρα πάλι βλέπουμε ότι η οικονομική ανισότητα, η μεγάλη απόκληση που υπάρχει στα εισοδήματα επωφελεί μόνο τους ε, έχοντες καθότι αυτοί μπορούν να αγοράσουν το μεγαλύτερο τμήμα ε, έγκυου ιδιοκτησίας. Βάσει λοιπόν όσο μας είπε μόλις ο Τζόναθαν, θα πρέπει να θέσουμε κάποια πολύ θεμελιώδη ερώτηματα για το κατά πόσο η κατανομή υγεών είναι η βέλτιστη για την ε, ε, λειτουργία της ιστορικής αγοράς. τότε λοιπόν την κατανομή στην διαφάνεια, βλέπουμε πόσο μεγάλη είναι η συγκέντρωση σήμερα στην Ευρώπη. Υπολογίσαμε βάσει των στοιχείων των δεδομένων της Eurostat ότι η συγκέντρωση είναι ως εξής. Μόνο 1% ε, ε, των ε, αγροκτημάτων ελέγχει το 20% της γης, 3% ελέγχει το 5% και μόνο 80% ελέγχει το 14,5% των γεών. Άρα λοιπόν δεν είναι δημοκρατική αυτή η διανομή και αυτό δημιουργεί διάφορα προβλήματα και ανισότητες στην γεωργία που τις ε, αναλύουμε στην μελέτη μας. Ουσιαστικά είναι δραματική η απώλεια των μικρών αγροκτημάτων. Μεταξύ 2003 και 2010 έπεσε κατά 25% ο αριθμός των αγροκτημάτων κάτω από 10 εκτάρια. Έτσι δεν υπάρχουν ευκαιρίες, θέσεις απασχόλησης, ε, επίπεδο φιλοδοξίας. Ε, δημιουργείται περιβαλλοντική ζημιά διάβρωση χάνουν ένα μεγάλο τμήμα της βιοπικιλότητας και επίσης δεν υπάρχει ανεξαρτησία και ασφάλεια σε ό,τι αφορά το τρόφιμα. Γιατί επιλέγεται πιο πολύ το μοντέλο των εξαγωγών. Και επίσης ε, υπάρχει και κάποια, κάποιες ε, μακροπρόθεσμες απειλές σε ό,τι αφορά για παράδειγμα ε, την γονιμότητα κάποιων ε, επιχειρήσεων γιατί ε, είναι πιο πιθανόν να φτωχεύσουν αυτές οι μεγάλες επιχειρήσεις. Επίσης και σε ό,τι αφορά την συσσόρευση χρεών και ενδεχόμενο σκάσιμο της φούσκας αυτής το αποτέλεσμα λοιπόν είναι μια κατάσταση της Ευρώπης χωρίς άμυνες, έτσι το αποκαλούμε. Δεν υπάρχει ένα σύστημα έγκυρης προειδοποίησης για να, κατα... για να εποπτεύει το σύστημα α, γεωργικής καλλιεργίας στην Ευρώπη και έτσι η έκταση και η πρόσβαση στα στοιχεία για την ε, παρακολούθηση της εφαρπαγής στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι επαρκής. ζητείτε να δημιουργηθεί ένα παρατηρητήριο για τις ευρωπαϊκές γέες. Πέρα από το τεχνικό κτηματολόγιο θα σε λέγει αυτό το παρατηρητήριο στοιχεία δεκαετούς περίοδου για κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των γεωκτημόνων, τις σχέσεις που έχουν με τις γεές και την εκμετάλλευση των γεών και θα περιλαμβάνει ενδεχομένω και κάποια βρελοντικά κριτήρια. Και πιστεύουμε λοιπόν ότι αυτό θα αποτελούσε ένα σημαντικό βήμα για να αναπτυχθεί ένα πανευρωπαϊκό, μια πανευρωπαϊκή βάση δεδομένων για τις ε, γεές στην Ευρώπη σήμερα. Κατά δεύτερον, η Ευρώπη είναι χωρί άμυνε γιατί είναι περιορισμένοι, Μάλλον είναι υπάρχουν ακόμα περιορισμοί στην μεταφορά κεφαλαίων και στις συστάσεις πολιτικής που έχουμε κάνει στη μελέτη μας. Θα δείτε ότι περιλαμβάνουμε διάφορες προτάσεις προκειμένου τα κάτι μέλη να αναπτύξουν και να συντονίσουν τους περιορισμούς που χρειάζεται για να αντιμετωπίζετε το, πρόβλημα της υφαρπαγής πιο αποτελεσματικά. θέση αυτή βασίζεται σε άλλες εκθέσεις που καταδεικνύουν πραγματικά ότι δεν έχουμε αρκετές ρυθμίσεις όσον αφορά την έγκυο διεκτησία. Βάσει ποιο κριτηρίων λοιπόν μπορούμε να βασιστούμε. Έχουμε κάποιες ε, κατευθυντήρες γραμμές όσον αφορά την έγκυο διεκτησία από τη ΦΑΟ που εγκρίθηκαν το 2012. Αναφέρονται οι κατευθύνσεις αυτές γραμμές στις ε, σχέσεις που υπάρχουν μεταξύ κρατών μελών και διεθνών οργανισμών όπως η ΦΑΟ και οι σε αυτές γραμμές για την διοκτησία γης έχουν ως στόχο να προστατεύσουν την έγκυο διοκτησία τουλάχιστον στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προβλέπεται μια διαβούλευση με τον τοπικό πληθυσμό, η διαφάνεια, το γενικό δημόσιο συμφέρον, καθώς ε, λαμβάνεται υπόψη και το τμήμα εκείνων των πληθυσμών το οποίο είναι πιο δεν έχει τόσο μεγάλη πρόσβαση στην έγκυο διοκτησία. Το τμήμα εκείνο το οποίο είναι πιο περιθωριοποιημένο. Δεν υπάρχουν ξεκάθαρες αρμοδιότητες ανάμεσα στα κράτη-μέλη και του ε, θεσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά το ζήτημα αυτό τη εγκύου διοκτησία. Ζητούμε λοιπόν από του Ευρωπαϊκού θεσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τα κράτη-μέλη να αναλάβουν ο καθένα τι ευθύνε του και προτείνουμε κάποια μέσα τα οποία θα μπορούσαν να εγκριθούν συστάσεις και προτάσει ουσιαστικά. Μία σύσταση έχει να κάνει με τη θέσπιση πολιτικών προτεραιοτήτων όσον αφορά την ιδιοκτησία γη. Επίση, το να καταφέρουμε να λάβουμε υπόψη μα τις τομεακές πολιτικέ Ευρωπαϊκή Ένωση το ζήτημα της ιδιοκτησίας γης. Κατά αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να προβλέψουμε δεσμευτικές ή υποχρεωτικές, υποχρεωτικά μέτρα. Προτείνουμε επίσης μία σειρά μέτρων τα οποία είναι ιδιαίτερα ενδιαφέροντα και τα οποία θα μπορούσαν ε, να χρησιμοποιηθούν για να μην έχουμε τέτοια συγκέντρωση ιδιοκτησία γη. Κάνουμε επίση και κάποιε συστάσει στο τέλο τη έκθεση, προκειμένου να χρησιμοποιήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο κάποια από τα εναλλακτικά μέτρα τα οποία προτείνουμε. Ο συνδυασμό λοιπόν των μέτρων αυτών ενδεχομένω να έχει πολύ θετικέ ε, επιδράσει. Καταρχάς, να έχουμε μια καλύτερη κατανομή των πληρωμών, έτσι ώστε πραγματικά να ευνοηθούν οι μικρότεροι παραγωγοί, να υπάρχει ένα το όριο όσον αφορά τις ενισχύσεις. Νομίζω ότι είναι παράλογο από ένα σημείο και μετά να πετάμε, να σπαταλούμε κατά αυτόν τον τρόπο δημόσιους πόρους, ιδίως στις πιο πλούσιες και μεγάλες γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Νομίζω ότι θα πρέπει επίσης να ξαναδούμε τον ορισμό του ενεργού γεωργού, γεωκτήμονα και να ξαναδούμε επίση τα ανώτατα όρια τα οποία έχουν τεθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν επιτρέπουν σε ορισμένου μικρού ενεργού καλλιεργητέ να έχουν πρόσβαση σε άμεσε ενισχύσει. Στα πλαίσια τη αναθεώρηση του προπολογισμού του 2017 θα μπορούσαν να γίνουν κάποιε επικοδομητικέ αλλαγέ στο καθεστώ τη ιδιοκτησία γη και επίση στην επόμενη περίοδο αναθεώρηση κοινή ζωρική πολιτική από το 2020 και μετά θα μπορούσαν να γίνουν οι απαραίτητε τροποποιήσει. Ολοκληρώνοντας, η έκθεση αυτή ευνοεί την έγκριση της κατάλληλης νομοθεσίας από τα κράτη-μέλη και γι' αυτό το λόγο θα ήταν καλό το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να καταδείξει μια κάποια ευελιξία και να επιτρέψει στα κράτη-μέλη να κάνουν τις απαραίτητες τροποποιήσεις και μεταρρυθμίσεις για να εγκρίνουν νέες νομοθεσίες και να υπάρχουν κάποιε βέλτιστε πρακτικέ μεταξύ κρατών μελών. Τι έχουμε εντοπίσει αυτέ τι βέλτιστε πρακτικέ και τι παραθέτουμε στην έκθεση αυτή. Τα βασικά διακυβεύματα λοιπόν είναι καταρχά να δούμε ότι η έγκυο ιδιοκτησία και το σχετικό καθεστώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε κοινοτικό και εγχώριο επίπεδο παρουσιάζει κάποια προβλήματα. Θα πρέπει να θετηθούν μέτρα για να θεραπευτούν τα προβλήματα αυτά και θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι η γη, η διοκτησία γης δεν μπορεί απλώς να αποτελεί προϊόν το οποίο θα θεσπίζεται στα πλαίσια μόνο τη ιστορική αγοράς, δεν είναι μόνο οικονομικό προϊόν, αλλά είναι ένα αγαθό το οποίο έχει έντονες κοινωνικές και πολιτιστικές πτυχέ. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ για την πολύ ενδιαφέρουσα αυτή παρουσίαση. Είμαι σίγουρος ότι οι συνάδελφοι έχουν πολλές ερωτήσεις να θέσουν. Ή δυνατόν να ξεκινήσω εγώ. Και καταρχάς να σας συγχαρώ. Η παρουσίαση ήταν πολύ ενδιαφέρουσα, πολύ κατατοπιστική. Απλώς να σας ρωτήσω, οι πηγές σας ποιες ακριβώς ήταν, από πού αντλήσατε όλες αυτές τις πληροφορίες. γιατί καταλαβαίνετε ότι τα όσα μας είπατε βαρύνουν και όλες πολιτικά έχουν μια πολύ έντονη πολιτική διάσταση. Συνεπώς σε τι βασιστήκατε, ποιες είναι οι πηγές σας. Δεύτερο ερώτημα. Το ζήτημα των μέσων που πρέπει να χρησιμοποιηθούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να μεταρρυθμιστεί το σύστημα εγγύου διοκτησίας. Ποια μέσα μπορεί να χρησιμοποιήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και ποια μέσα μπορεί να χρησιμοποιήσουν τα κράτη-μέλη όταν δρούμε μονομένα. Συμφωνώ με τα όσα είπατε ότι όντως ε, η γη δεν μπορεί να αποτελέσει απλό οικονομικό προϊόν αντικείμενο αγοράς και πώληση στα πλαίσια μιας εσωτερικής αγοράς. Συμφωνώ με αυτό. Αλλά στην πράξη τι μπορούμε να κάνουμε με κάποιες βασικές αρχές, με κάποια βασικά νομοθετήματα τα οποία ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά την έγκυη ιδιοκτησία. Ξέρετε ότι το ζήτημα αυτό απασχολεί πολλά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως και το ζήτημα της συγκέντρωσης της ιδιοκτησίας γης. Και κάτι ακόμα, Έχετε το λόγο, παρακαλώ. Πολύ σας ευχαριστώ. Μεγάλη τιμή που μιλάω πρώτη-πρώτη. Θα ήθελα και εγώ από δική μου πλευρά να ευχαριστήσω πάρα πολύ του συζητητέ για την παρουσίαση τη μελέτη. Έχω συχνά την αίσθηση ότι ξεχνάμε σε διάφορε περιστάσει ε, τα μικρά πράγματα τα οποία όμως έχουν μεγάλο αντικτύπο στην Ευρώπη. Η αναδιανομή των γεών λοιπόν, το είπατε ξεκάθαρα, είναι κάτι το οποίο υφέρπει στα κρατημέλη, αλλά το οποίο επηρεάζει με αρνητικό τρόπο και πολύ μαζικά την κοινωνία μας. Δεν βρίσκω τίποτε το θετικό στο ότι όλο και πιο λίγα άτομα ελέγχουν και κατέχουν μεγαλύτερες εκτάσεις γεών. Είναι λοιπόν αρνητικό αυτή η μονομερής διαχείριση των γεών. Μιλήσατε για τις άμεσες ε, πληρωμές. Θα ήθελα να μου πείτε πώς εκτιμάτε το θέμα ότι οι άμεσε ε, πληρωμές αυτέ δίνονται αποκλειστικά στους ιδιοκτήτε. Δηλαδή, με το σύστημα αυτό στην Ευρωπαϊκή Ένωση ουσιαστικά ε, παρατρύνουμε και δίνουμε κίνητρα σε αυτή την αγορά των γεών από κάποιους λίγους ε, γεωκτήμονες. Και τελικά δεν ωφελούνται αυτοί που θα έπρεπε να ωφελούνται. Πώς λοιπόν ε, αξιολογείται την κατάσταση αυτή και πόσα χρήματα τελικά πηγαίνουν στα στην τσέπη του καλλιεργητή και πόσα καταλήγουν στην τσέπη του επενδυτή. Αυτό θα ήθελα να μου πείτε, ο κύριος Χόισλινγκ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσίαση της μελέτης. Διαπιστώνουμε λοιπόν στο πλαίσιο αυτό ότι το land grabbing, αυτή η φαρπαγή καλλιεργειών είναι για πολλούς από εμά κάτι που συμβαίνει στην Ασία, στην Αφρική, αλλά δεν μας απασχολεί στην Ευρώπη. Νομίζω ότι με τη μελέτη αυτή αποδεικνύεται ότι θα πρέπει να μπει αυτό στην ημερήσια διάταξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το θέμα της διανομής ε, των ε, γεωργικών εκτάσεων και διοκτησιών στην Ευρώπη αποτελεί ένα μεγάλο θέμα. Και βλέπουμε από τη μελέτη αυτή ότι χρειάζεται κατεπηγόντως να αναλάβουμε δράση. Η βάση δεδομένων είναι ισχνή. Έχετε δίκιο ότι αυτό που χρειάζεται σε πρώτη φάση είναι μια διαφάνεια. Σε όλα τα κράτη-μέλη θα πρέπει να διευκρινίζεται ε, ποιοι έχουν τη γη προκειμένου να υπάρξει τουλάχιστον μια καταγραφή του φαινόμενου της συγκέντρωσης των γεών. Δεύτερο ερώτημα, πώς θα αντιδράσουμε και αυτό το περιγράψατε. Υπάρχουν ε, μεγάλες ε, εταιρείε κεφαλαίων που αποκτούν τέτοιε γεές ε, ως επένδυση. Πώς μπορούμε λοιπόν να αντιμετωπίσουμε το φαινόμενο αυτό, να μένει δηλαδή η γη στα χέρια όσων την καλλιεργούν και την εκμεταλλεύονται πραγματικά. Πώς μπορούμε λοιπόν να παρέμβουμε στο σημείο αυτό. Μιλήσατε για την Ουγγαρία και την Πολωνία συγκεκριμένα και είπατε το πώς ε, γίνονται αγορές μέσω ε, εταιριών ε, ψεύτικων. Μέσω εικονικών εταιριών. Πώς μπορούμε λοιπόν να αντιμετωπίσουμε για το φαινόμενο αυτό. Εδώ λοιπόν πιστεύω ότι υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη καλύτερη ενημέρωση. Τι γίνεται, πού, πόσο απειλητικά είναι τα φαινόμενα αυτά και πώς μπορούμε πολιτικά να αντιδράσουμε. Θέσατε το ερώτημα του κατά πόσον πρόκειται για αρμοδιότητα εθνικών κρατών μελών ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιστεύω ότι είναι αρμοδιότητα και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί αν εμείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση ε, δίνουμε κίνητρα και επιταχύνουμε τη διαδικασία αυτή θα έπρεπε ίσω να ξανασκεφτούμε το θέμα των άμεσων πληρωμών. Θυμάμαι μια συζήτηση όπου είχε προτείνει, α, ε, είχε προτείνει όριο ανάμεσα 300.000 ευρώ, ε, άλλοι προτείνανε 150.000 ευρώ. Θα πρέπει ίσως να το ξανακοιτάξουμε αυτό το θέμα. Μήπως με τις άμεσες επιδοτήσεις ε, αν δεν βάλουμε κάποιο ανώτατο όριο, ουσιαστικά προωθούμε τη μεγαλύτερη συγκέντρωση στα χέρια των επενδυτών. Αυτή η συζήτηση λοιπόν θα πρέπει να ξαναγίνει. Πιστεύω και θα ήθελα και οι άλλε ομάδε να το βάλουν αυτό στη μερίσια διάταξη, να συζητήσουμε μήπω το θέμα αυτό θα έπρεπε να μα οδηγήσει σε μια έκθεση πρωτοβουλία, προκειμένου να μπει σε, ως πολιτική προτεραιότητα το θέμα αυτό. Η ομάδα μας σίγουρα θα ήταν υπέρ. Γιατί ε, αυτή η μελέτη περιλαμβάνει τόσα πολλά δεδομένα που πιστεύω ότι θα μπορούσαν να αρκέσουν για μια έκθεση πρωτοβουλία. Πολύ σα ευχαριστώ. Πάνη Πόσου Χόιμπους. Κύριος Η κυρία Χόιμπου. Ευχαριστώ πολύ. Χάρηκα πολύ με τη μελέτη αυτή, με την έρευνα αυτή, γιατί παρουσιάσατε το πρόβλημα από πολλέ οπτικές γωνίε. Και προσπαθήσατε να καταλήξετε και σε μια σύσταση για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρουσιάσατε και τις δράσει δράσεις που θα μπορούσαμε να αναλάβουμε από τη ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί φυσικά λόγω της ελεύθερης διακίνησης ε, των γεών Τη ιδιοκτησία δηλαδή, των Υγεών Δεν έχει μεγάλα περιθώρια η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά πραγματικά μα δώσατε κάποιε εναλλακτικέ για το ποιε δράσει θα μπορούσαμε να αναλάβουμε. Πολύ σα ευχαριστούμε λοιπόν. Θα πρέπει να βρούμε το κατάλληλο πλαίσιο λοιπόν εδώ για την ε, αποκοινού διαμόρφωση του ζήτηματο στην Ευρώπη. Έχω πάρα πολλέ ερωτήσει, αλλά α περιοριστώ σε δυο τρει καλύτερα. Επανέρχομαι λοιπόν ε, στο θέμα της διαμόρφωσης της πολιτικής. Μιλήσατε για τις κατευθυντήριες γραμμές. Ερωτώ, αυτές οι εθελούσιες, οι εθελοντικές κατευθυντήριες γραμμές ε, είναι γνωστές, είναι ενημερωμένα το κοινό για αυτές. Στα κράτη-μέλη εφαρμόζονται. 125 κράτη έχουν προσυπογράψει αυτέ τι εκατευθυντήριε γραμμέ, αλλά δεν σημαίνει ότι εφαρμόζονται φυσικά σε αυτά τα 125 κράτη. Θα ήθελα λοιπόν να μα πείτε αν έχετε κοιτάξει κατά πόσον υπάρχει εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών αυτών στι ευρωπαϊκέ χώρε. Ύστερα, μιλήσατε για τη βάση δεδομένων σε ό,τι αφορά τον πίνακα γεών. Και μιλάμε για 4,3 εκατομμύρια εκτάρια γεών έχει συνυπολογιστεί και η Ρωσία και η Ουκρανία. Αλλά μας είπατε ότι λείπουν και πολλά δεδομένα. Ήθελα να ρωτήσω, έχετε κοιτάξει το χρονικό παράγοντα. Μετά την χρηματοπιστωτική κρίση στην Ευρώπη έχουν αυξηθεί οι αγοραπολισίες γεών ή είναι σταθερά τα πράγματα τα τελευταία 10-15 χρόνια. Και μια τελευταία ερώτηση τώρα, επιτρέψτε μου. Το είπατε και στην παρουσίασή σας για το ότι 3% των εταιριών ελέγχουν 50% των ε, γεών των αγροπημάτων στην Ευρώπη. Πρόκειται για ομίλους, γεωργικούς, ευρωπαϊκούς επενδυτές. Ποια είναι η σύσταση δηλαδή του 3% αυτού που κατέχουν το 50% των εκτάσεων. Έχετε στοιχεία ή κυρίως εκτιμήσεις κάνετε. Και με χαρά θα ακούσω και τις ερωτήσεις των υπόλοιπων συναδέλφων. Ευχαριστώ. Ο κύριο Ντές. Σας ευχαριστώ για τις παρουσιάσεις σας αυτές. Θα πρέπει να το κοιτάξουμε το θέμα αυτό πιο επισταμένος. Ο σοσιαλισμός όμως στην Ευρώπη ήταν εκείνος που πήρε από τους αγρότες την ίδια του στη γη. Και σήμερα ακόμα ε, υποκείμεθα σε αυτές τις συνέπειες του σοσιαλισμού. Στη Γερμανία υπάρχει πολύ αυστηρός νόμος για την μεταβίβαση διακτησίας των γεών και παρόλα αυτά αυτός ο πολύ αυστηρός νόμος δεν μπορεί να αποτρέψει συγκέντρωση εκτάσεων. Για παράδειγμα, στην, στο κατηδίο Μέκλεμουγκ Πάμερ. Και θα πρέπει να κοιτάξουμε το θέμα από διάφορες οπτικές γωνίες. Μου προκαλεί πραγματικά τρόμο το γεγονός ότι είπατε ότι στη Ρουμανία ε, οι επιχειρήσεις μέχρι 5.000 ευρώ δεν λαμβάνουν ε, καμία πληρωμή. Αυτό πρέπει να είναι αναμφίβολα νομοθεσία της Ρουμανίας, της ρουμανικής κυβέρνησης, γιατί στην Ευρώπη σίγουρα δίνουμε ε, χρήματα στις μικρές επιχειρήσεις. Και στη Γερμανία επιδοτούνται ιδιαίτερα οι μικρές ε, καλλιέργειες μέχρι 30 εκτάρια. Μέχρι 46 εκτάρια πρέπει να τουλάχιστον 2.000 ευρώ επιπλέον επιδοτήματα. Στην Βαβαρία, στην Τουρκία εξετάσαμε ε, αγροκτήματα με 600 αγελάδες, 3.500 ε, εκτάρια. Αλλά αυτά α, ανήκουν σε 261 ιδιοκτήτες. Ανά άτομο, ούτε τρεις αγελάδες δεν βγαίνουν. Γιατί πρόκειται λοιπόν για μια κύριη νομική κατάσκευη, ένα συνεταιρισμό. Πρόκειται για 261 ιδιοκτήτε που κατέχουν από κοινού του 800 αγελάδε. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να γίνει μια διαφορετική αξιολόγηση. Και ξέρω ότι αν εισαγαγούμε ανώτατα όρια, το συζητήσαμε επισταμένω και στην γεωργική μεταρρυθμίση, και εμεί στη Βαβαρία αποφασίσαμε να υπάρχουν τέτοια ανώτατα όρια. Αλλά αυτό ξέρετε δεν αποτελεί κανένα πρόβλημα για τους μεγάλους ε, ομίλους, γιατί μπορεί να σπάσουν μια ιδιοκτησία σε πολλές ε, μικρότερες. Άρα είναι περιορισμένος ο αντίκτυπος του μέτρου του ανώτατου ορίου. Εγώ είμαι κατά της ε, ίδρυσης νέων υπηρεσιών σε ό,τι αφορά το παρατηρείο. Αλλά φαντάζομαι ότι η Γενική Διεύθυνση Άγκρη θα μπορούσε να δημιουργήσει μια υπηρεσία παρακολούθηση του ζητήματος και βλέπουμε ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα μπορούσαμε να καταλήξουμε σε μια απόφαση προκειμένου τουλάχιστον τα κάτι μέλη να αναφέρουν τι γίνεται στην επικρατεία τους για να είμαστε ενήμεροι και να μπορούμε να παρακολουθούμε με καλύτερο τρόπο πώς κινούνται οι μεγάλοι όμιλοι, τα μεγάλα κεφάλαια. Γιατί αυτό ασφαλώς δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα μιας σωστής και καλής ανάπτυξης στην Ευρώπη. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα θα ήθελα να εξετάσουμε εδώ το πρόβλημα στη Ρουμανία, γιατί δεν είμαι πεπισμένος ότι εξαιρούνται ή αποκλείονται από τις ενισχύσεις οι μικρές εκμεταλλεύσεις. Πρέπει να το επανεξετάσουμε. Τώρα κύριε Ομπούντα, στη συνέχεια τώρα κύριε Σταραμπέλα. Ευχαριστώ πρόεδρε που μου δίνετε το λόγο και μου δίνετε την ευκαιρία να μιλήσω για τις ε, άμεσες πληρωμές ε, στη Ρουμανία. Οι μικρές, ε, τα μικρά, οι μικρές καλλιέργειας λαμβάνουν επιδοτήσεις στη Ρουμανία. Δεν τίποτα πιο τίποτα τέτοιο θέμα. Ωστόσο, οι ομιλητές μίλησαν για τη συγκέντρωση των εκτάσεων στα χέρια των μεγάλων επενδυτών. Αυτό λοιπόν αληθεύει. Και δεν μιλάμε για ε, εταιρείε μόνο από το Λίβανο, αλλά από όλο τον κόσμο. Το μεγάλο λοιπόν πρόβλημα είναι το πού καταλήγουν τελικά τα χρήματα. Τα χρήματα δεν πηγαίνουν στους μικρούς ε, καλλιεργητές πλέον. Σε αυτούς που θα έπρεπε να υποφελούνται, αλλά τελικά καταλήγουν στα χέρια των μεγάλων επενδυτών. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να εξετάσουμε τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πώς θα πρέπει να εξελιχθούν για τα θέματα της ε, αγοράς εκτάσεων. Όσο δύσκολο και αν είναι το θέμα αυτό, θα πρέπει να το ρυθμίσουμε στο εγγύς μέλλον. Ιδάλλως, υπονομεύουμε τις ίδιες μας τις πολιτικές. Δίνουμε στον κόσμο α, χρήματα, επιδοτήσεις για να αντιτηρηθούν θεωρητικά οι μικρές καλλιέργειες, αλλά ουσιαστικά τα χρήματα καταλήγουν στις τσέπες άλλων. Κύριε θα πρέπει πραγματικά ως κοινοβούλιο να λάβουμε άμεσο δράση. Εντάξει. Εάν κατάλαβα λοιπόν, οι μικροί γεωργοί λαμβάνουν ενίσχυση. Ωραία. Ο κύριος Σταραμπέλα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Είναι σημαντικό να απαντήσω μετά τον κύριο Ντέ, γιατί παρότι κόπηκε στα δύο η Ευρώπη μετά το 1945, ο κομμουνισμός πράγματι έκανε την εφαρπαγή των γεών, όμω, ε, η σημερινή πραγματικότητα είναι η επανενωμένη δημοκρατική Ευρώπη. Και αυτό ο ανεξέλεγκτο καπιταλισμό ε, προβαίνει στην εφαρπαγή σε όλο τον, τον κόσμο μάλλον, και στην Αφρική και στην Ασία και στην Ευρώπη. Δεν ξεφεύγουμε αυτόν τον κανόνα. Το πρόβλημα υπάρχει και στη Ρουμανία, γιατί σίγουρα έχει θα αυξηθεί μάλλον τρομερά η παραγωγή με τα επόμενα χρόνια, γιατί έχει πολύ γόνιμες γέες και θα αυξηθεί και η παραγωγικότητα. Και έτσι σίγουρα θα είναι η χαρά του επενδυτή. Και στο, σε βάρος λοιπόν και εννοείται των μικρών καλλιεργητών. Το βλέπουμε και στη χώρα μου, στο Βέλγιο, ότι όταν σταματούν οι μικροί καλλιεργητές, κάποιες φορές ε, υφαρπάσσονται υγιές από τους γείτονε, όμως όλα είναι και περισσότερο από μεγάλες αγροοικονομικές επιχειρήσεις και το ερώτημα που θέλω να θέσω είναι πολύ απλό. Και ο κύριος το έθιξε. Έχουμε καλούς μηχανισμούς ανακατανομής των επιδοτήσεων. Θυμάμαι και αυτό το ποσό των 200.000 ευρώ με σταδιακή κατάργηση, το οποίο είχε καταψηφιστεί για δύο ψήφους στην Ολομέλεια. Γιατί υπήρχαν αιτήματα για μεγαλύτερη κατανομή. Όμως βλέπουμε ότι και πάλι ο καπιταλισμός αυτός ο ανεξέλεγκτος, ε, εκεί μας έχει οδηγήσει, δεν θέλουμε καμία ρύθμιση, κανέναν έλεγχο. Ε, θα σταματήσουν ε, οι επιδοτήσεις για τη ζάχαρη, για το γάλα σε δύο χρόνια. Επομένω υπάρχει η τεράστια πτυτικότητα που είναι ο εχθρός του γεωργικού επενδυτή Μήπως θα πρέπει να έχουμε και αντικυκλικές ε, επιδοτήσεις, γιατί για παράδειγμα η τιμή του τόνου ε, ε σιτηρών είναι 240 ευρώ, δεν έχει κανένα νόημα να έχει κάποιος επιπλέον επιδοτήσεις. Κάτι το οποίο συνέβαινε το 2010. Δεν έχει νόημα δηλαδή να έχουμε ευρωπαϊκές επιδοτήσεις ε, σε σημαντικές αγορές. Όμως από την άλλη για παράδειγμα στο γάλα μπορούμε να τους ε, ε, στηρίξουμε. Αντικυκλικές λοιπόν επιδοτήσεις και επανασύνδεση ε, των επιδοτήσεων και αυτό δεν είναι βρισιά. Αν δείτε τι συμβαίνει στον κόσμο, στις μεγάλες χώρες παραγωγούς, Βραζιλία, ΙΠΑ, που συνδέουν τις επιδοτήσεις τους. Εμείς είμαστε μοναδικοί που κάνουμε το αντίθετο και δημιουργούμε δυσκολίες για το μικρό καλλιεργητή. Ευχαριστώ πολύ. Δεν έχω θέσει ακόμα χρονικό όριο για τις παρεμβάσεις, γιατί έχουμε ακόμα χρόνο. Όμως, από εδώ και πέρα, θα ήθελα να σας παρακαλέσω να, να μείνατε στα δύο λεπτά στις παρεμβάσεις σας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, λέει ο Θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτό που έθιξε και η κυρία Κέι. Μίλησε για παράνομες ε, αγοραπολισίες στην Πολωνία. Πράγματι, στην Πολωνία υπάρχει νόμος που προστατεύει την ε, πρόσβαση στην πολωνική γη απέναντι στους ξένους, στους αλλοδαπούς. Παρά αυτό το νόμο όμως, το έχετε δει και εσείς, ότι υπάρχουν πολλοί ξένοι φορείς που αγοράζουν γη στη χώρα μου μέσω διαφόρων τεχνασμάτων. Μιλήσατε για 200.000 εκτάρια και είπατε ότι αυτό το φαινόμενο αφορά κυρίως τη Δυτική Πολωνία. Εάν υπάρχει δυνατότητα, θα ήθελα να μας πείτε ποια είναι η πηγή των δεδομένων που σας επέτρεψε να καταλήξετε σε αυτό το συμπέρασμα. Κάθε χρόνο το Πολωνικό Κοινοβούλιο ασχολείται με αυτό το ζήτημα και ε, το Υπουργείο Εξωτερικών παρουσιάζει έκθεση για τις ε, αγορές γης από αλλοδαπούς και πρέπει να πω ότι κάθε φορά που ακούω αυτή την έκθεση ο Υπουργός ε, το μόνο που ανέφερε ήταν κάποιες εκατοντάδες εκτάρια και εσείς ξαφνικά μιλάτε για 200.000 εκτάρια. Θα ήθελα λοιπόν να μου πείτε ποια δεδομένα σας οδήγησαν σε αυτό το συμπέρασμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εξέτασα την μελέτη και είδα ότι δεν έχετε αριθμητικά στοιχεία για την Κροατία. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να με διαφωτίσετε. Θα θέλαμε κάποια αριθμητικά στοιχεία για την Κροατία που είναι εδώ και δύο χρόνια μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το θέμα λοιπόν που τίθεται και τα ερωτήματα που θέσατε είναι θέματα που εμπίπτουν στον τομέα αρμοδιοτήτων των ε, κυβερνήσεων. Μιλάμε για τη χρήση των γεωργικών εκτάσεων. Αυτές λοιπόν οι κυβερνήσεις είναι αρμόδιες για τον καθορισμό της πολιτικής αυτής. Ε, στην Κροατία μετά το σοσιαλιστικό καθεστώς ε, βλέπουμε ότι η υπάρχουν ε, μικρές εκμεταλλεύσεις που είναι στην ε, ιδιοκτησία των μικρών γεωκτημόνων. Το πρόβλημα όμως που αντιμετωπίζουμε είναι ότι αυτές οι καλλιέργειες δεν ήταν βιώσιμες, πολύ απλά. Δεν μπορούσαν να επιζήσουν τα οικονομικά προβλήματα δε, τα οποία αντιμετωπίσαμε, ήταν η βάση για την κατανομή των ε, εκτάσεων μετά την πολιτική αλλαγή. Και μεγάλες εταιρείε πλέον έχουν θηγατρικές και στην Κροατία. Και έτσι παρατηρούμε το εξή φαινόμενο. Ότι μία θηγατρική, για παράδειγμα, έχει, όλα τα, έχει στην της όλα τα ζώα και η άλλη έχει μόνο την ε, γεωργική έκταση. Και έτσι λοιπόν ε, δίδονται για παράδειγμα εκτάσεις στην εταιρεία που έχει μόνο στην διεκτησία της τα ζώα. Θα πρέπει λοιπόν από ευρωπαϊκή πλευρά να ορίσουμε κατά πόσον η κοινή γεωργική πολιτική όντω ωφελεί τι μικρέ επιχειρήσει, τι μικρέ εκμεταλλεύσει. Αν λοιπόν αυτό επιθυμούμε, θα πρέπει να βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη, γιατί αν δεν υπάρχουν αυτοί οι μικροκαλλιεργητέ, αυτοί οι μικροειδιοκτήτε, δεν θα υπήρχε ζωή στην Ήπεθρο και η Ήπεθρος πραγματικά θα νεκρονόταν. Ο αγρότης λοιπόν, ο καλλιεργητής, δεν είναι μόνο υπεύθυνο για τη διατήρηση της βιοπικιλότητας, ε, της ε, προστασίας του περιβάλλοντος, όχι. Είναι αυτός που βάζει το φαγητό στο τραπέζι και αυτός που κρατάει ζωντανό το χωριό. Γι' αυτό λοιπόν, αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη σε ό,τι αφορά την κατανομή των εκτάσεων. Στην Κροατία λοιπόν βλέπουμε ότι οι μικρέ οικογενειακέ εκμεταλλεύσει ουσιαστικά πλέον δεν είναι βιώσιμε. Γιατί δεν του επιτρέπουμε να ζήσουν, του κόβουμε το οξυγόνο. Θα πρέπει λοιπόν να του δώσουμε μεγαλύτερο περιθώριο. Το θέμα λοιπόν είναι στην Κροατία κατά πόσον υπάρχει μεγάλε αλλοδαπέ ή και οι μεδαπέ ε, Επιχειρήσει και όμιλοι, γιατί εξαφανίζονται λοιπόν με τον τρόπο αυτό οι μικρέ επιχειρήσεις. Ευχαριστώ. Κυρία Μπίλερ. Μίλες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ και για την μελέτη η οποία αποτελεί ένα σημείο εκείνη. Είναι εδώ και 35 χρόνια είμαι αγρότης και πάντα υπήρχε μια κάποια αλλαγή των δομών και αυτό είναι και απαραίτητο. Πριν από 13 χρόνια είχαμε 18 εκτάρια, τώρα έχουμε 70 εκτάρια. Μια οικογένεια στο τελική ανάλυση πρέπει και αυτή. Α, δεν με ακούτε. No, no translation. Υπάρχει όμω, Υπάρχει όμως, υπάρχει. Eine Familie muss auch Geld verdienen. Οι οικογένειε λοιπόν, οι αγροτικέ οικογένειε θα πρέπει λοιπόν να κερδίζουν χρήματα στην τελική ανάλυση και γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να αναπτύσσονται. Άρα σε πολλού τομεί υπάρχει ανάγκη διόρθωση. υπάρχουν πολλοί νόμοι στη Γερμανία για τι αγροτικέ εκτάσει, πολλοί αυστηροί νόμοι, οι οποίοι όμω δεν φτάνουν για να αποκλειστούν οι ανισότητε και οι ανισορροπίε. Είναι λοιπόν σημαντικό το γεγονός ότι με, το, με τη μελέτη αυτή κάνουμε μία αρχή, μία κίνηση. Αλλά σύμφωνα με την πρόταση του κυρίου Ντες, πως στη Γενική Διεύθυνση Άγκρη θα μπορούσαν να, να συλλέγονται δεδομένα από όλα τα κράτη-μέλη για να υπάρχει μια βάση δεδομένων. Χωρίς μια τέτοια βάση δεδομένων, χωρίς μια επακριβή παρακολούθηση του τι συμβαίνει σε κάθε κράτος μέλος, δεν θα μπορέσουμε να παρέμβουμε. Στην Γερμανία ενισχύονται οι μικρές επιχειρήσεις σε άλλες χώρες, ε, ε, υπάρχουν συνδεδεμένες ε, επιδοτήσεις. Δεν υπάρχει λοιπόν αυτή η κυνηγερική πολιτική. Και παρόλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντική η διάσταση προστασίας των ιδιωτών ή ταξιτών. Και θα πρέπει όντως να δούμε τι έκταση γης είναι στα χέρια των ίδιων των καλλιεργητών. Θα πρέπει λοιπόν αυτό να το ξέρουμε, προκειμένου να μπορέσουμε να προβούμε σε εξαγωγή συμπερασμάτων. Όταν λοιπόν ολοκληρώσουμε τη διαδικασία αυτή, όταν μπορούμε να μιλήσουμε για πραγματικά γεγονότα, τότε θα μπορέσουμε να αποφασίσουμε αν χρειάζεται δράση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Κύριε Πρόεδρε, Χαίρομαι πάρα πολύ που μπορώ και συμμετέχω στη συζήτηση αυτή. Θεωρώ ότι πραγματικά αντιμετωπίσουμε ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα και θα πρέπει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να το λύσουμε αυτό το οποίο βλέπουμε στο μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ότι θα έχουμε όλο και μεγαλύτερες ανισορροπίες όσον αφορά την διοκτησία γης και θα πλήττεται όλο και περισσότερο γεωργικός αγροτικός πληθυσμός. Νομίζω ότι θα όλο και περισσότερο προς μια πολύ μεγάλη συγκέντρωση ιδιοκτησία γης. Πρέπει να αντιταχθούμε και να καταπολεμήσουμε αυτή την τάση. Και νομίζω ότι βλέπουμε όλο και περισσότερο μια περίμωση των υπαίθριων περιοχών. Πρέπει λοιπόν να καταφέρουμε να διατηρήσουμε ζωντανή την ύπεθρο αν χάσουμε τις θέσεις απασχόλησης στην ύπεθρο εξαιτίας της συγκέντρωσης ιδιοκτησίας γης, τότε πολύ φοβάμαι ότι θα έχουμε περισσότερες γεωργικές εκτάσεις μεν, αλλά πολύ λιγότερο ενεργό αγροτικό πληθυσμό. Για ποιο λόγο έχουμε αυτή τη συγκέντρωση γης. Ξέρετε ότι ε, οι περισσότεροι μικροκαλλιεργητές όταν αποχωρίζονται βασικά το αγρόκτημά τους χρειάζονται ουσιαστικά χρήματα. Το πουλάνε προκειμένου να καταφέρουν να κερδίσουν κάποια χρήματα. Και κατά αυτόν τον τρόπο εκχωρώντας γη, ο καλλιεργητής θα έπρεπε αντί να δίνει τη γη του σε μεγάλες πολυεθνικές επιχειρήσεις να μπορεί να τις εκχωρεί, να τις παραχωρεί σε νέους μικρούς καλλιεργητές. Να πω δύο πράγματα όσον αφορά τη μελέτη αυτή. Δεν ξέρω αν είδατε καθόλου στα πλαίσια της έρευνάς σας τη δυνατότητα που υπάρχει όσον αφορά την οικοδόμηση των γεωργικών αυτών ε, γεών. Ξέρετε ότι και αυτό αποτελεί ένα πρόβλημα. Βλέπουμε όλο και περισσότερο ότι χάνονται γεωργικές εκτάσεις ακριβώς επειδή οικοδομούνται στα περίχωρα πόλεων. Δεν ξέρω αν επίσης ε, <clears throat> εξετάσετε το ζήτημα των δασικών εκτάσεων το γεγονός ότι ε, πολλές φορές ορισμένες καλλιεργήσιμες εκτάσεις που εγκαταλείπονται καλύπτουν τελικά από βλάστηση, από δέντρα και δεν μπορούν να ανακτηθούν από τους καλλιεργητές στη συνέχεια. Ευχαριστούμε. Κοιτάξτε, και εγώ όταν ε, σκέφτομαι το ζήτημα αυτό της συγκέντρωσης, ε, της ιδιοκτησίας γης, Αναρωτιέμαι αν τελικά υπάρχει ένα ευρωπαϊκό μοντέλο όσον αφορά την ιδιοκτησία γη στην Ευρώπη και θα μπορούσαμε ουσιαστικά να υιοθετήσουμε και ένα παγκόσμιο τέτοιο μοντέλο. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τους δύο προσκεκλισμένους μας. Οι πληροφορίες μας δώσαν είναι πολύ σημαντικές. Κατά την άποψή μου το πρόβλημα είναι πολύ σημαντικό. Θα έπρεπε λοιπόν, να μη τι άλλο, να συντάξουμε μια έκθεση πρωτοβουλία για αυτό το ζήτημα. Ξέρετε ότι στην Πολωνία αντιμετωπίζουμε ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα. Τα τελευταία χρόνια στην Πολωνία φοβόμαστε όλο και περισσότερο εξαιτία τη διεύρυνση αυτή τη πρακτική Από την 1η Ιανουαρίου του 2016 μήπως θα μα αγοράσουν, θα μας εξαγοράσουν μαζικά οι ξένοι. Αυτό είναι ο φόβος ε, που τρέφουν πάρα πολλοί Πολωνοί. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο οικονομικό, είναι ένα σημαντικότατο κοινωνικό πρόβλημα. Πέρα από τις γενικές έρευνες που έχουν γίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά την αλλαγή της διάρθρωσης της διοκτησίας γης, πέρα από αυτό λοιπόν θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και τα ιδιαίτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ανατολικές χώρες της Ευρώπης. Ξέρετε ότι στα ανατολικά της Ευρώπης η γη κοστίζει λιγότερο από ό,τι στη Δυτική Ευρώπη και αυτό από μόνο του προσελκύει πολλούς ξένους επενδυτές. Οι τοπικοί όμως πληθυσμοί θα επιθυμούσαν να διατηρήσουν την ιδιοκτησία γης, να διατηρήσουν τις καλλιεργίες τους και να διασφαλίσουν τελικά ότι αυτό το εθνικό περιουσιακό στοιχείο θα διασωθεί. Θα ήθελα λοιπόν να συντάξουμε μια έκθεση πρωτοβουλίας κύριε Πρόεδρε και έχω και ένα ερώτημα ακόμα και ολοκληρώνω. Θα ήθελα και εγώ να γνωρίζω ποιες είναι οι πηγές που χρησιμοποίησαν οι συντάκτες της μελέτης. Βάσει ποιο πληροφοριών καταλήξατε στα στατιστικά δεδομένα μας παρουσιάσετε όσον αφορά την κατάσταση στην Πολωνία. Ο κύριος ε, Ανταγωγιά έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω τους ε, δύο υπεύθυνους της μελέτης αυτής. Η παρουσίασή τους καταδεικνύει τα αποτελέσματα της δικής μας κοινοτικής πολιτικής όσον αφορά την γεωργία και τους περιορισμούς, τα όρια της πολιτικής αυτής. Και συμφωνώ και εγώ ότι θα είναι πολύ σημαντικό πολύ γρήγορα να συντάξουν μια έκθεση πρωτοβουλίας για μια μελλοντική μεταρρύθμιση της κοινή διορικής πολιτικής μετά το 2020, χωρίς να περιμένουμε την ενδιάμεση αξιολόγηση. Τα όσα ακούσαμε αντιστοιχούν σε ένα πάρα πολύ σημαντικό πρόβλημα. Το γεγονός ότι η γη όντως αποτελεί περιουσιακό στοιχείο, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μια σφαιρική προσέγγιση όσον αφορά το δημόσιο αυτό περιουσιακό στοιχείο. Ακούσαμε πάρα πολλά πράγματα για τη διακύμαση των τιμών, για την πτυτικότητα των τιμών, για το γεγονός ότι ε, χάνουμε θέσεις απασχόλησης, το γεγονός ότι η κοινή γεωργική πολιτική δεν ανταποκρίνεται στα αγρονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η Πεθρός. Πρέπει λοιπόν να δούμε αν όντω η πολιτική που ακολουθούμε είναι καλή, αν όντω είναι κατάλληλη, αν είναι πλέον αποτελεσματική. Κάθε φορά που εφαρμόζουμε λοιπόν μια δημόσια πολιτική η οποία χρησιμοποιεί ως βασικό τη στοιχείο της ε, αποσυνδεδεμένες ενισχύσεις, ε, τότε δεν είναι τυχαίο το ότι έρχονται πάρα πολλοί ξένοι επενδυτές οι οποίοι θέλουν να αγοράσουν τις γέες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καταλαβαίνετε ότι επίσης μέσω της πολιτικής των ορίων που έχουμε στις άμεσες ενισχύσεις και πάλι προσελκύουμε πολλούς ξένους δυνατούς επενδυτές οι οποίοι έρχονται για να εξαγοράσουν ευρωπαϊκή γη. Και ξέρετε ότι ε, βασικό τους μέλημα είναι τα οικονομικά του συμφέροντα, πώς θα καταφέρουν να πτύξουν περισσότερο τις δραστηριότητές τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και βλέπουμε ότι παρόλα αυτά, μόλον ότι βλέπουμε τόσο αρνητικά αποτελέσματα από την κοινή γεωργική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνεχίζουμε και προωθούμε την πολιτική αυτή. Θα ήθελα και εγώ να γνωρίζω ποιες είναι οι πηγές σας. Νομίζω ότι πραγματικά αν βασιστούμε στις πηγές αυτές, θα πρέπει να επιναρρυθμίσουμε κάπως και την πολιτική την οποία ακολουθούμε και τη σχέση γης και απασχόλησης. Δεν ξέρω αν οι ενισχύσεις αυτές που δίνουμε έχουμε όντω κάποια θετική επίπτωση στην απασχόληση στην Ήπεθρο. Οι δημόσιες πολιτικές που ακολουθούμε ουσιαστικά κατέστησαν κάποιες περιοχές ακόμα πιο ευάλωτες. Ε, εγκατελείφθηκαν πάρα πολλά τμήματα της υπαίθρου και συγκεντρώθηκαν κάποια, κάποιες αγροτικές εκμεταλλεύσεις σε πολύ συγκεκριμένα σημεία μόνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό νομίζω ότι πρέπει να μας απασχολήσει και νομίζω ότι βασιζόμενοι στα στοιχεία σας αυτά θα καταφέρουμε να καταρτήσουμε μια νέα πολιτική μετά το 2020. Ευχαριστώ μας δίνεται πολύ τροφή για σκέψη και είναι μια πολύ καλή πρωτοβουλία. Ωστόσο, όπως είπαν και οι συνάδελφοι, πρέπει να εξετάσουμε τις πηγές των στοιχείων που μας παρουσιάσατε. Και γιατί το λέω αυτό. Γιατί στις ε, παραπομπές ε, της ε, παρουσίασής σας, εσείς παραθέσατε ένα άρθρο εφημερίδας που είναι ουσιαστικά συνέντευξη του Υπουργού Γεωργίας. θα ήταν σκόπιμο τα, οι αρχές που ασχολούνται με αυτά τα ζητήματα στα κράτη-μέλη ή μάλλον εσείς θα πρέπει να είστε σε επαφή με αυτά τα Ινστιτούτα, αυτούς τους θεσμούς, αυτές τις αρχές. Γιατί όταν παραπέμπεται σε άρθρα εφημερίδων, τότε εύκολα μπορεί να ξεφύγει και να εκτροχιαστεί η συζήτηση. Όπως είπε και ο κύριος Ντες, μπορεί τελικά να δημιουργηθεί σύγχυση και να θεωρούμε ότι ε, οι γεωργοί στη Ρουμανία δεν παίρνουν επιδοτήσεις, αλλά όλοι παίρνουν από, από έκταση 0,3 εκταρίων. Δεν υπάρχει διαφοροποίηση ε, μεταξύ των ε, Ρουμανών ή άλλων γεωργών. Και τώρα έχουμε το νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης για την Ήπεθρο. Οι μικροί καλλιεργητές παίρνουν μάλιστα τέτοιες επιδοτήσεις συμπληρωματικές για να τους ενθαρρύνουμε να δώσουν τα προϊόντα τους στην αγορά. Θα ήθελα να ακούσω την γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για αυτή την έκθεση. Υπάρχουν εδώ εκπρόσωποι της Κομισιόν. Θα ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρον να ακούσουμε και την γνώμη της Επιτροπής λοιπόν. Επίσης, νομίζω ότι στη μελέτη σας θα ήταν σημαντικό να μας πείτε ποιες θα ήταν πιθανές λύσεις από στατιστικής άποψης. Πώς μπορούμε να αποτρέψουμε τους ξένους να εφαρπάξουν τη γη μας. Τι πρέπει να κάνουμε, να επιτρέψουμε στους νέους γεωργούς να αγοράσουν τη γη που θέλουν. Νομίζω λοιπόν ότι τα κράτη-μέλη πρέπει να έχουν αυξημένο ρόλο σε αυτό το τομέα. Νομίζω ότι ε, είναι όλα θετικά αυτά που αναφέρουμε είμαι υπέρ μια τέτοια ε, έκθεση πρωτοβουλία, αλλά πρέπει να δούμε και τα στοιχεία που προκύπτουν. Ο κ. Νταντά, ευχαριστώ. Η μελέτη είναι ενδιαφέρουσα και λάβαμε γνώση ε, σήμερα το πρωί, επομένω χρειαζόμαστε χρόνο να την μελετήσουμε σε βάθο. Το ζήτημα αυτό είναι πιο περίπλοκο από ό,τι έχει αναφερθεί μέχρι τώρα. Για τι πράγμα μιλάμε. Μιλάμε για εκμετάλλευση της γης ή για την κτίση, την ιδιοκτησία τη γη γιατί η χρήση γης αποτελεί αρμοδιότητα των μελών. Και σε κάθε κράτος μέλος υπάρχουν ε, διαφορετικοί νόμοι και κανονισμοί. Αυτό ισχύει και στη Γαλλία. γιατί ε, μετά τον δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ήταν ιδιοκτήτε οι Γεωργοί σε ποσοστό 75% ενώ σήμερα είναι πολύ πολύ μικρότερο. Δεν ε, μπορούμε να πούμε ότι διάφορες προσπάθειες που είχαν καταβληθεί ε, στέθηκαν με επιτυχία. Όμως και πάλι ε, μια καλλιέργεια μπορεί να έχει πολλές μορφές. Ποιος είναι ο κάτοχος του μετοχικού κεφαλαίου, για παράδειγμα. Είναι 4, 5, 6 μέλη μιας οικογένειας είναι μια καπιταλιστική εταιρεία που δεν έχει καμία σχέση με την γεωργική εκμετάλλευση. Πρέπει να τα διαφοροποιήσουμε αυτά. Και μετά υπάρχει και μια άλλη έννοια Εγώ έρχομαι από μια ορεινή περιοχή. Ε, το γεγονό ότι υπάρχει χαμηλή παραγωγικότητα ή δυνατότητα καλλιέργεια για μόνο τρει μήνε το χρόνο, αυτό σημαίνει ότι είχαν μεγάλε εκτάσει ε, στα βουνά οι, οι καλλιεργητέ οικογένειε και μικρότερε εκτάσει στι παιδιάδε. Αυτό το σημαίνει πρέπει να του δούμε σαν μεγάλου καλλιεργητέ. Όχι, πρέπει να τα εξετάσουμε σε μεγαλύτερο βάθο τα πράγματα στι μελέτε, να διαφοροποιήσουμε και το νομικό πλαίσιο και το ε, κοινωνικό πλαίσιο και την χρήση της γης. Και όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, πώς εξετάζουμε και το ζήτημα ε, του αστικού πλαισίου. Εμείς έχουμε 100 νομούς. Τους τελευταί, τα, τελευταία χρόνια έχουμε χάσει ε, έκταση αντίστοιχη ενός τέτοιου νομού ε, εξαιτίας της ε, αστικοποίησης. Και αυτό επειδή υπάρχουν και διαφορετικές πιέσεις που ασκούνται και πρέπει να το εξετάσουμε συνολικά το ζήτημα. Και όχι μόνο σε ό,τι αφορά την ε, κατανομή των επιδετήσεων της ΚΑΠ, που είναι ένας παράγοντας που μας επηρεάζει μεταξύ άλλων. Ευχαριστώ. Κύριε Ντόρφμαν, ευχαριστώ Πρόεδρε. Η συζήτηση την οποία κάνουμε μου προκαλεί μια κάποια έκπληξη, πρέπει να ομολογήσω. Κοιτώντα τι ε, βασικέ ε, εξελίξει και τι τα βασικά κινήματα στην Ευρώπη, είναι λίγο δύσκολο να μιλάμε για land grabbing. Είναι λίγο επικίνδυνο, πιστεύω. Υπάρχουν κάποιε διαδικασίε οι οποίε ενδεχομένω να υπάρχουν στη διαδικασία αυτή. αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις οικογενειακών επιχειρήσεων που απλά μεγαλώνουν. Στην Ιταλία, για παράδειγμα, πολλοί νέοι και στη Ρουμανία ε, το τελευταίο καιρό έχουν αγοράσει νέες εκτάσεις ε, και είναι πλέον σήμερα γεωργοί. Είναι κακό αυτό. Είναι αυτό η φαρπαγή γεών. Εάν ε, αναφέρουμε ότι είναι αυτά αρνητικά ζητήματα, τι να πω, και η δυνατότητα ελεύθερη εγκατάσταση και η δυνατότητα ελεύθερη μετακίνηση είναι δύο βασικέ αρχέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη. Στην Ουγγαρία, για παράδειγμα, που υπάρχουν αυτά τα pocket contracts, αυτό γίνεται γιατί δεν επιτρέπονται άλλε μορφέ αγορά εκτάσεων. Αυτό που είναι πολύ ενδιαφέρον ωστόσο στην μελέτη αυτή και έχουν δει και απόλυτα οι υπεύθυνοι που την κατήρθησαν ότι η δική μας πολιτική, η γεωργική πολιτική θα πρέπει να εξετάσει πιο επισταμένα τα φαινόμενα συγκέντρωσης. Να δούμε δηλαδή ποιος λαμβάνει, ποιος είναι αυτό το 3%, από ποιον την αποτελεί αυτό το 3% που κατέχει το 50% των εκτάσεων. Έχει σχέση με τους πραγματικούς καλλιεργητές. Και να πούμε και το εξή στο σημερινό χρηματοπιστωτικό κόσμο είναι δύσκολο να υπάρχει βέβαιη απόδοση, σίγουρη απόδοση. Ή επιχειρήσεις που έχουν μεγάλο κεφάλαιο αναζητούν όλο και πιο πολύ σίγουρες αποδόσεις. Και με τη δική μας πολιτική δυστυχώς συμβάλλουμε προς την κατεύθυνση αυτή. Γιατί η απόδοση της καλλιέργειας γης είναι κάτι σίγουρο ως εισόδημα. Αυτό δεν μπορεί να αποτελεί καλή πολιτική για τις οικογενειακές επιχειρήσεις. Θα ήθελα να σχολιάσω εν συντομία τα όσα υπόθηκαν. Για παράδειγμα στην Πολωνία έχουμε περιπτώσεις όπου ε, Ολλανδοί υπήκοοι έχουν αγοράσει 100-150 εκτάρια. Δεν ζουν αυτοί οι άνθρωποι στην... Ε, ή μάλλον, συγγνώμη, ε, ζουν αυτοί οι άνθρωποι στην Πολωνία, καλλιεργούν τη γη τους και δεν υπάρχει εκεί πέρα πρόβλημα. Γιατί πραγματικά ζουν και εργάζονται στην Πολωνία. Δεν το θεωρούμε κάτι αρνητικό, αντιθέτω είναι μια θετική συγκέντρωση. Όμω για μα η φαρπαγή γεωργική γη συμβαίνει όταν το πρόσωπο δεν ε, δραστηριοποιείται πραγματικά σε αυτή την εκμετάλλευση. Κύριο Γιάννη. Σα ευχαριστώ, Πρόεδρε. Νομίζω ότι είναι σημαντικό το θέμα τη ιδιοκτησία. γιατί έχει να κάνει και με την πολιτική μας και με την κατοικοποίηση όλων, αλλά νομίζω ότι μια ευρεία κατανομή της συντεκτησίας σταθεροποιεί την κοινωνία και το αντίθετο φυσικά προκαλεί ανισότητες, ανισορροπίες και αποσταθεροποίηση. Θα πρέπει λοιπόν ε, να κοιτάξουμε επισταμένο στο θέμα της κατανομής της συντεκτησίας ε, εκτάσεων. Να βάλουμε λίγο νερό στο κρασί μας επίσης. Οι άμεσες πληρωμές δεν μπορεί να τις κατηγορούμε για όλα. Στη Γερμανία δεν είναι καν σημαντικό μέτρο. Γιατί δεν επηρεάζουν ιδιαίτερα την παραγωγή. Αυτό ω υπόδειξη. Τρία πράγματα έχω σημειώσει να σα αναφέρω. Καταρχά, χαίρομαι που έχουμε την μελέτη αυτή και τη χρειαζόμαστε μεγαλύτερη και όλο και πιο πολύ ανάλυση τη κατάσταση. Και κάποιε αρχέ για την ανάλυση. Βλέπουμε στη σελίδα 33 ότι υπάρχουν σημαντικές διαφορές Μιλάμε για 5% των ε, δικαιούχων, 0,8%. Θα πρέπει λοιπόν να κάνουμε αναλύσει να αναπτύξουμε και ένα σύστημα για τα κράτη-μέλη που θα κάνει τα καθήκοντα λίγο συγκρίσιμα, γιατί υποθέτω στην παρούσα φάση δεν είναι συγκρίσιμα τα πράγματα. Για να χρησιμοποιήσουμε τη Γενική Γραμματεία για την ανάλυση αυτή, εδώ συμφωνώ. Επίσης, να συμφωνήσουμε τι είναι μικρό, τι είναι μεγάλο, ποιος είναι ο ρόλος ε, ε, του ανταγωνισμού και τέλος, τι θα πρέπει και τι θέλουμε να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο αυτό. Επαναλαμβάνω, είναι σημαντική η διεκτησία, είναι μια εντική μορφή διεκτησίας η γη και γι' αυτό θα πρέπει να μας απασχολήσει πιο πολύ. Και αν ε, θέλετε να κάνουμε έκθεση πρωτοβουλία θα ήμουν σύμφωνο για να έχουμε πιο πολύ ευκαιρία να το συζητήσουμε στην Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σα ευχαριστώ πολύ καταρχά για αυτό το έγγραφο, τη μελέτη αυτή που μα δίνει κάποια στατιστικά δεδομένα τα οποία συγκλίνουν και με τι πληροφορίε που είχαμε εμεί οι ίδιοι στην Πολωνία. Να επανέλθω τώρα στο πρόβλημα της συγκέντρωσης γεωργικών γεών. Ποιος υποφελείται από αυτό το φαινόμενο. Για ποιο λόγο βλέπουμε το φαινόμενο αυτό να πτήσεται όλο και περισσότερο. Όταν κάναμε την επίσκεψη μελέτη στην Φιλανδία, ενημερωθήκαμε εκεί πέρα με κάποια αριθμητικά δεδομένα που μας έδωσε το Υπουργείο της Φιλανδίας. Το 1990 είχαμε περίπου 130.000 γεωργικές εκμεταλλεύσεις, εκ των οποίων οι περισσότερες ήταν 17 εκτάρια, με περίπου συνολικά έσοδα και κέρδη ένα δισεκατομμύριο. Τώρα βλέπουμε ότι έχει μειωθεί κατά το ίμιση και η έκταση αυτών των εκτάσεων, αλλά και στα έσοδα των γεωργών. Βλέπουμε λοιπόν ότι το φαινόμενο της συγκέντρωσης των γεών οδηγεί τελικά και σε μείωση των γεωργικών κερδών. Για ποιο λόγο δηλαδή να υφίσταται το φαινόμενο αυτό, για ποιο λόγο να υπάρχει έντονη αυτή συγκέντρωση γεωργικών γεών, όταν τελικά αυτό δεν συμβάλλει στην ανάπτυξη της όταν αυτό δεν συμβάλλει καν στην ανάπτυξη της κερδοφορίας. Νομίζω ότι ανταυτού αυτό που βλέπουμε είναι ότι μειώνεται η γεωργική παραγωγή μέσω τη συγκέντρωση γεωργικών γεών. Ειλικρινά δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο η κοινή γεωργική πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση επιτρέπει αυτή την ε, καλπάζουσα αύξηση τη συγκέντρωση γεών. Και επίση είδαμε ότι υπάρχουν και πολύ αρνητικέ περιβαλλοντικέ επιπτώσει από αυτό το φαινόμενο. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να βαθύνουμε περισσότερο στο ζήτημα και να μας απασχολήσει το ερώτημα της μελλοντική τελικά γεωργικής πολιτικής που θα πρέπει να εγκρίνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι είδους γεωργία θέλουμε για το μέλλον. Πρέπει να δημιουργήσουμε ευνοϊκές συνθήκες για τους μικρούς καλλιεργητές και τις μικρές οικογενειακές γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Και κάτι ακόμα κύριε Πρόεδρε και ολοκληρώνω αντιμετωπίζουμε ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα, το οποίο έχει να κάνει με την ανισότητα του ανταγωνισμού στα εσωτερικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε δύο διαφορετικές Ευρώπες. Μία Ευρώπη δύο ταχυτήτων όσον αφορά την γεωργία. Μία πολύ πλούσια Ευρώπη στα δυτικά και μία πολύ φτωχή Ευρώπη στα ανατολικά της Υπήρου. Οφείλουμε συνεπώς να βρούμε λύσεις και σε αυτό το πρόβλημα, προκειμένου να καταφέρουμε να προστατεύσουμε τους γεωργούς από την Ανατολική Ευρώπη. Διαφορετικά καταλαβαίνετε ότι ανοίξουμε περισσότερο την αγορά γη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν θα έχουν κανένα κέρδος πλέον αυτοί οι μικροί καλλιεργητές, ιδίως στην Ανατολική Ευρώπη. Ευχαριστώ. Ένα σύντομο σχόλιο. το μέγεθος της λεγόμενης μικρής εκμετάλλευσης ποικίλει βεβαίως και εδώ πρέπει να το εξετάσουμε αυτό το θέμα. Нека да от там, че изследването наистина е много важно, тъй като земеделието... Ευχαριστώ, πρόεδρε. Και θα ήθελα να ξεκινήσω λέγοντας ότι η μελέτη αυτή είναι εξαιρετικά σημαντική, γιατί η γεωργία και οι γεωργικές εκτάσεις αποτελούν την ε, βάση όλων των δράσεων από πλευράς του Υπουργείου Γεωργίας. Και ποια, ε, ποια είναι η θεσμική, ποια είναι οι θεσμή που θα πρέπει να προστατεύσουν τις ε, γεωργικές εκτάσεις. Οι επενδυτέ θέλουν να αγοράζουν εκτάσει για να έχουν απόδοση. Τι γίνεται όμω με τι εκτάσει που έχουν υποστεί διάβρωση. Συμφωνώ λοιπόν για τους λόγους αυτούς ότι χρειαζόμαστε μια έκθεση πρωτοβουλίας προκειμένου να γίνουν κάποιες προτάσεις και ίσως θα έπρεπε να καθιερωθεί ένα σύστημα ανταλλαγής και σύγκρισης βέλτιστων πρακτικών. Στην Βουλγαρία υπάρχει πολιτική σε ό,τι αφορά τα διαβρωμένα εδάφη, τις διαβρωμένες αγροτικές εκτάσεις. Η καλλιέργεια δε από διάφορα άτομα σημαίνει μεγαλύτερη απασχόληση γιατί το έδαφος είναι το καθημερινό ψωμί, ξέρετε, ο άρτος επιούσιος. Και συνεπάγεται και κοινωνική ασφάλεια για τον κόσμο στην Ήπετρο. Σταθερότητα. Προσπαθούμε λοιπόν να συγκέντρωση, να πετύχουμε συγκέντρωση της γεωργίας για να υπάρχει μεγαλύτερη εξασφάλιση και στην περίπτωση αυτή βλέπουμε ότι καταλείπονται οι ορεινές περιοχές για παράδειγμα. Χρειαζόμαστε μια δίκαιη πολιτική και θα πρέπει να συγκρίνουμε λοιπόν ποια είναι τα αποτελέσματα και οι συνέπειε των άμεσων επιδοτήσεων. Γιατί είναι καλή πρόθεση ασφαλώς να επιδοτηθούν οι μικροί καλλιεργητές, οι μικροί εκμεταλλευτές, αλλά τελικά αυτό ωφελεί τους μεγάλους επενδυτές. Γιατί τελικά αυτοί τσεπώνουν τελικά τα χρήματα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μιλήσα για τα εικονικά αυτά, τις εικονικές αυτές ε, συμβάσεις ε, στην Ουγγαρία, για τις εικονικές εταιρείε μίλησε ο κύριος Τες. Για τα pocket contracts αυτά, αυτές τις εικονικές συμβάσεις, οφείλονται, ακούσαμε, στις ε, διατάξεις της νομοθεσίας. Υπάρχουν σχετικοί νόμοι στην Δανία, στην Γαλλία και επί της βάσης αυτής ε, ε, αναλάβουμε στην, αναλάβαμε νομική δράση στην Ουγγαρία και βλέπουμε λοιπόν ότι προκαλούνται προβλήματα. Φυσικά, ζητούμε και αγωνιζόμαστε για μεγαλύτερη δικαιοσύνη και οι Αυστριακοί γεωκτήμονες αγοράζουν μέσω εικονικών εταιριών εκτάσεις χωρίς να κατοικούν στην Ουγγαρία. Θα ήθελα λοιπόν να διευκρινίσω ότι αυτά που συμβαίνουν και αυτά που οργανώζονται σωστά στην Δανία και στην ε, Γαλλία είναι αυτός ο νόμος για την μεταβίβαση διοκτησίας ε, εκτάσεων. Αν κατατίσαμε λοιπόν ένα παρόμοιο νόμο σχέδιο προκειμένου να δημοσιοποιηθεί μια δίκαιη κατάσταση και στην Βαρία. Ευχαριστώ κύριε Σκακαλινόφσκι. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ε, η μελέτη που μας ε, και είναι πολύ καλή και θα θέλω να σας ευχαριστήσω. Μιλήσατε για τις ανησυχητικές ε, τάσεις που παρατηρούνται σε ό,τι αφορά τη συγκέντρωση γης. Επίσης, δώσατε και κάποια παραδείγματα κερδοσκοπικών αγορών. Αυτό αφορά κυρίως την Ανατολική Ευρώπη, την Πολωνία, την Ουγγαρία, τη Ρουμανία Μιλήσατε ακόμα και για ενδιαμέσους που έχουν την πολωνική υπηκότητα, έχουν το δικαίωμα να αγοράσουν γη στην Πολωνία και έτσι γίνονται εικονικοί ιδιοκτήτες. Ποιο είναι το πρόβλημα λοιπόν, ότι παίρνουν χρηματοδότηση ε, ξένων επενδυτών και μετά από μία σύντομη χρονική περίοδο οι ξένοι επενδυτές θα υφαρπάξουν τη γη. Στα στατιστικά λοιπόν στοιχεία δεν περνάει και δεν καταγράφεται αυτή η ξένη διεκτησία. Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, έχουμε κάποιους ε, νόμους στο δίκαιό μας, καθώς και έναν, ε, μια υπηρεσία που διαχειρίζεται την αγοραπολισία γης και έχουμε και συγκεκριμένο κατόφλι σε ό,τι αφορά τη γεωργική εκμετάλλευση στην Πολωνία. Πάνω από 300 εκτάρια αυτή η υπηρεσία έχει δικαίωμα ε, προτεραιότητας ό,τι φορά την αγορά αυτή τη γης. Όταν κάποιος αγοράζει αυτή την, αγορά, την ε, γη θα πρέπει να πρόκειται για φυσικό πρόσωπο. Τώρα, αν είναι μια εταιρεία που αγοράζει τη γη, Εκεί πέρα υπάρχουν ε, ασάφειες και κενά στην νομοθεσία. Πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε αυτά τα προβλήματα, να βρούμε λύσεις για να θέσουμε τέλος ε, στην κερδοσκοπία στη γη. Γιατί υπάρχει πολύ σημαντικό πρόβλημα σήμερα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θεματοφύλακα των ε, Ευρωπαϊκών Συνθήκων, μας διαβεβαιώνει ότι Αυτά τα νομοσχέδια που έχουν ως στόχο την προστασία των γεών, αυτά τα νομοσχέδια λοιπόν έρχονται σε αντίθεση με το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Εμείς ως Κοινοβούλιο πρέπει να ε, ασχοληθούμε το συντομότερο δυνατόν με αυτό το θέμα και να καλέσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αλλάξει την προσέγγιση της, γιατί αυτή τη στιγμή ενεργεί υπέρ των κερδοσκόπων. Σας ευχαριστώ και πάλι για τη μελέτη. Ευχαριστώ πολύ. Να δώσουμε τώρα το λόγο στη Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ Πρόεδρε που μας δίνει τη δυνατότητα να σχολιάσουμε την τομή αυτή τη μελέτη. Πρώτα απ' όλα το θέμα που εξετάζουμε που είναι ιδιαίτερα ευρύτερο για, ε, για τα δικαιώματα χρήση γη και μεταβίβασή του. Όλα αυτά είναι ιδιαίτερα περίπλοκα και πρέπει να τα μελετήσουμε περαιτέρω πριν καταλήξουμε στι συμπεράσματα, γιατί είναι και θέμα αρμοδιότητα των κρατών μελών και υπάρχουν σημαντικά κενά στα στοιχεία. Χαιρετίζουμε τι προσπάθειε ε, αναζήτηση νέων στοιχείων για να προσιωθεί αυτή η συζήτηση. Ωστόσο, η μελέτη μπλέκει διαφορετικέ διαφορετικές χωρί να δίνει μια καλή και εύρωστη κατανόηση ε, του αντιτύπου τη υφαρπαγή, ενώ ε, ερμηνεύεται μεροληπτικά ε, το φαινόμενο ε, με συγκεκριμένα στερεότυπα σε ό,τι αφορά την δομή και την εκπαιδευτική της χρήσης γης. Έχουμε και αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που είχε ως ε, στόχο να εξετάσει τον αντίκτυπο των άμεσων ενισχύσεων ε, στις διαρθρωτικέ μεταρρυθμίσεις. Και εδώ είχαμε επιτάχυνση της διαρθρωτική μεταρρύθμισης λόγω της αποσύνδεσης, το οποίο ήταν κάτι ε, αναμενόμενο και επιθυμητό. Και αυτό αξιοποιείται ως απόδειξη και στοιχείο για το τι συμβαίνει στην εφαρπαγή γεών. Για την ίδια την εφαρπαγή, η, η έκθεση αναφέρει ότι υπάρχει ε, διάσταση απόψεως ό,τι αφορά τον ορισμό και δεν υπάρχει μία και μόνο ε, άποψη. Όμως περιπλέκει συνεχώς ε, την έννοια της εφαρπαγή γεών που δεν ορίζεται πουθενά με τη συγκέντρωση, τις διαφορετικέ μεταρρυθμίσεις, ακόμα και τις άμεσες ξένες επενδύσει στη γεωργία. Δεν λέμε ότι δεν είναι σοβαρά αυτά τα ζητήματα, μάλιστα σε δύο εξολογήσεις αντικτύπου και στο Health Check και στην πρόσφατη μεταρρύθμιση της CAP υπάρχει πολύ εκτεταμένη ανάλυση και αναλύσεις που έχουμε αναθέσει σε εξωτερικούς ε, φορείς για, ακριβώς για την διασύνδεση μεταξύ άμεσων ενισχύσεων και αγοράς ε, γης. Όμως, δεν υπάρχουν στοιχεία συγκεκριμένα για το πεδίο εφαρμογή και την κλίμακα αυτού του φαινομένου. Τα στοιχεία αναφέρουν σε έκταση 166.000 εκταρίων και σε πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις ε, στα κάποια κρατημέλη. Αυτό είναι η μεγαλύτερη απόδειξη ότι το θέμα είναι πολύ μικρό και αμεληταίο, γιατί αυτό είναι το 0,1% της συνολικής γεωργικής γης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως και να έχει, όσο και να το υποτιμούμε, το 0,1% με ό,τι και να το πολλαπλασιάσετε, με όποιο συντελεστή, πάλι μικρό ποσοστό θα έχετε. Επίσης, η ανάλυση της έκτασης της συγκέντρωσης γεωργικής γης εξετάζει μόνο τις εκμεταλλεύσεις άνω των 100 εκταρίων. Δεν εξηγεί γιατί υπάρχει αυτό το αυθαίρετο κατόφλι. Πολύ διαφορετικό για τα σιτηρά, ε, την κτηνοτροφία, εκτατική, όχι γεωργία, ε, μόνιμες καλλιέργειες όλα αυτά τι σύνδεση έχουν με το γενικό επιχείρημα. Το γενικό επιχείρημα λοιπόν ότι υπάρχει στενή διασύνδεση τη συγκέντρωση ε, υγιή και ε, ε, εκμετάλλευση δεν αναπτύσσεται. Δεν υπάρχει αναφορά στου διάφορου στους διάφορους παράγοντες που συνδέονται με την αλλαγή χρήση και δεν υπάρχει και αναφορά στο θεσμικό πλαίσιο και την χάραξη πολιτικής για την χρήση υγιής επιμέρους κρατημέλη έχουν πολύ διαφορετικές νομοθεσίες και για την μεταβίβαση γης και για την κληρονομιά και βλέπουμε ότι παρότι η γη είναι όπως είναι, η διοκτησία, ε, η ενοικίαση γης είναι από το 18% στα 20% στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ κατά μέσο όρο είναι 50%. Πιο συγκεκριμένα η ανάλυση κάποιες φορές περιπλέκει την ε, ε, κατανομή ε, πληρωμών ΚΑΠ με την εφαρπαγή γης, χωρίς να λαμβάνει υπόψη το γεγονός ότι η κατανομή των πληρωμών ΚΑΠ συνδέεται με την υφιστάμενη δομή και όχι το αντίστροφο. Το αν θα βασίσουμε τις επιδοτήσεις σε παρελθοντικές, προηγούμενες δηλαδή καλλιέργειες, παραγωγές όπως συνέβαινε πριν από 20 χρόνια ή στο ε, μέγεθος της έκτασης όπως συμβαίνει τώρα, πάντα θα υπάρχει άνεση κατανομή επιδοτήσεων, εκτός και αν έχουμε μια κατάσταση όπου κάθε γεωργός θα έχει την ίδια έκταση γης, το οποίο δεν είναι ρεαλιστικό και δεν πιστεύω ότι είναι και στέο. Τέλος, ό,τι αφορά τη διασύνδεση μεταξύ αγροτικών επιχειρήσεων, συγκέντρωση στην επιστημική αλυσίδα και εφαρπαγή γεών, δεν δίνονται στοιχεία. Και αυτό είναι ένα ε, τομέα που χρήζει περαιτέρω εξέταση, γιατί έχουμε πολύ ανάμεικτε εξελίξει σε διάφορα μέρη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Κλείνοντα, υπάρχουν και άλλα ζητήματα για την παραγωγικότητα, αγροτικός πληθυσμό, ε, φραγμή στην είσοδο, ε, στην αγορά και το καθεξής, ιδίως για τους νέους γεωργούς. Όμως, ιδιαίτερο ενδιαφέρον δείχνουν τα εξή στοιχεία. Πρώτα είχαμε τη διαφάνεια με τα πέντε ε, υφιστάμενα στοιχεία της ΚΑΠ. Μπορούμε επάπειρον να συζητήσουμε αν θα μπορούσαν ε, να ακολουθήσουμε διαφορετικό μείγμα και τι θα εφαρμόσουν τα κράτη-μέλη. Σύντομα θα έχουμε τα πρώτα αποτελέσματα, όμως αυτό είναι το σημείο εστίασης που μας δείχνει ποια είναι η κύρια προτεραιότητα. Χρήση γης και η αλλαγή χρήσης γης. Αυτό θα πρέπει να είναι το κύριο σημείο έμφασης της πολιτικής. Και υπάρχουν και δύο εναλλακτικέ στην πρόταση. Πρώτον, περιορισμοί στη μεταβίβαση κεφαλαίου προς άτομα, προς πρόσωπα. Η γη είναι ε, αμετάβλητο στοιχείο και γι' αυτό και ε, αποτελεί δύο τρίτα των περισσοκών στοιχείων της μεταρρύθμισης. Δηλαδή το θέμα είναι ότι αν εμείς από πλευράς δημόσιας παρέμβασης ε, εξετάζουμε και αντιμετωπίζουμε τις τα προβλήματα με, μετά την παρουσίασή τους ή εάν θα προσπαθήσουμε εκ των προτέρων να περιορίσουμε την μεταβίβαση κεφαλαίου και έτσι ε, αποτρέπουμε τα προβλήματα πριν δημιουργηθούν. Και το άλλο στοιχείο που ακούστηκε είναι οι αντικυκλικές επιδοτήσεις που έχουν χρησιμοποιηθεί εκτεταμένα στις ΕΠΑ και έχουμε δει τα αποτελέσματα. Σε ό,τι αφορά την κατανομή της ε, γης, τη συγκέντρωση της γης σε, στα δύο άκρα, έχουμε δει τη μεταβίβαση συγκεκριμένου βάρους σε, στους άλλους, γιατί οι γεωργοί ε, ασχολούνται μόνο με τη μεταβλητή του καιρού που δεν μπορούν να ελέγξουν και έχουμε δει και τα πτήσεμε στα αλλακτρομικά για παράδειγμα όπου με την αντικυκλική επιδότηση βλέπουμε ότι όσοι τη χρειάζονται παίρνουν λιγότερη στήριξη από ό,τι χρειάζονται. Θα είναι λοιπόν κεντρικό ζήτημα σε αυτή τη συζήτηση, όμως πρέπει να καταλήξουμε σε συγκεκριμένα συμπεράσματα. Για να το κάνουμε αυτό πρέπει να επισέλθουμε σε λεπτομέρειες και στο υπόβαθρο της κατάστασης. Γι' αυτό πιστεύουμε ότι σύντομα θα έχουμε στοιχεία για τη νέα διαρθρωτική μελέτη της Eurostat που θα μας επιτρέψει να λάβουμε υπόψη όλες τις αλλαγές που έγιναν ε, στην Ευρώπη και στην Ευρωπαϊκή Γεωργία τα τελευταία 10 χρόνια για να διευκρινίσουμε λίγο παραπάνω αυτά τα ζητήματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, μετά την παρέμβαση αυτή Νομίζω ότι πρέπει να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας προετοιμάσει ένα έγγραφο, ένα είδος πληροφόρησης για το ζήτημα αυτό συγκεκριμένα ή δυνατόν για το φθινόπωρο, έτσι ώστε να μπορέσουμε κι εμείς να καταλάβουμε καλύτερα τι συμβαίνει και ποια είναι τα επιχειρήματα τελικά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Λοιπόν, να ζητήσω τώρα από τους εμπειρογνώμονές μας να πάρουν το λόγο. Ας είστε σας παρακαλώ πολύ σύντομοι, μην περάσουμε τώρα σε άμεση αντιπαράθεση. Σας ευχαριστώ πολύ για όλες αυτές τις ερωτήσεις που υποβάλλατε. Πραγματικά ήταν πάρα πολύ θετικό το ότι είχαμε τέτοια ανταπόκριση στην έκθεση αυτή. Να ξεκινήσω με τις πηγές των πληροφοριών μας. Πολλοί το ρώτησαν αυτό. Προφανώς, στο τέλος της μελέτη θα δείτε όλη τη βιβλιογραφία και τις πηγές μας. Να αναφερθώ σε μερικές συγκεκριμένα πηγές που χρησιμοποίησαμε προκειμένου να καταφέρουμε να σας δείξουμε ποια είναι η κλίμακα της συγκέντρωσης και της υφαρπαγής γεών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Χρησιμοποίησαμε την έρευνα Factor Markets, μια έρευνα η οποία επιδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, σειρά έρευνων μάλιστα, και ιδιαίτερα χρησιμοποίησαμε την έρευνα από το 2012 όσον αφορά τον κανονισμό πώληση γεωργικών γεών και τον, τη σχετική έρευνα για τους κανονισμούς που διέπουν το εμπόριο των γεωργικών γεών σε διάφορα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, αντλήσαμε πληροφορίες από μια γνωμοδότηση ιδίας πρωτοβουλίας από την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινωνική Επιτροπή που έκανε μια έρευνα και αυτή για το land grabbing και νομίζω ότι θα ήταν πάρα πολύ καλό και εσείς ως Επιτροπή Γεωργίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να κάνετε μια μελέτη ιδίας πρωτοβουλίας. Το 2015 πάντως δημοσιεύθηκε η ε, έκθεση της ΕΟΚΕ, όπου παρουσιάζει το land grabbing, την υφαρπαγή και όνος απειλή για την Ευρωπαϊκή Ένωση και αναφέρεται στο ότι 200.000 εκτάρια από την Πολωνία έχουν περάσει σε ξένα χέρια. Από εκεί πήραμε λοιπόν αυτή την πληροφορία. Η τρίτη ε, σημαντικότερη πηγή πληροφοριών είναι ένα βιβλίο που δημοσίευσε το TNI το 2013 ζητήσαμε από 13 ε, ερευνητές εθνικό και τοπικό επίπεδο σε διάφορες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ανατολική και τη Δυτική Ευρώπη ε, περιβαλλοντικές οργανώσεις, οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κτηνοτροφικοί και γεωργική συνεταιρισμοί. Τους ζητήσαμε λοιπόν να κάνουν μια έρευνα επιτόπου και να επιλέξουν στοιχεία για κάθε χώρα ξεχωριστά. Παρουσιάσαμε τα στοιχεία αυτά τον Ιούνιο εκείνου του έτους και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σας εθαρρύνω λοιπόν να δείτε και τη μελέτη αυτή. Αυτά όσον αφορά τις πηγές μας. Ακούσαμε και μια ερώτηση για τη δυνατότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αναλάβει δράση προκειμένου να σταματήσει το φαινόμενο της αφαρπαγής γεών. Ως προς αυτό, θα έλεγα ότι το βασικό επιχείρημα που προωθεί η έκθεσή μα είναι ότι χρειάζεται καταρχάς σίγουρα δράση σε ευρύτερο ευρωπαϊκό επίπεδο για να σταματήσει αυτό το φαινόμενο γιατί μολονότι υπάρχουν κάποιες καλές βέλτιστες πρακτικές μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχουν πάλι πολύ μεγάλες διαφορές. Για παράδειγμα, στην Γαλλία το σύστημα διαρθρώνεται περισσότερο σε τοπικό περιφερειακό επίπεδο. Σε άλλες χώρες οι αποφάσεις λαμβάνονται σε πιο κεντρικό επίπεδο. Πάντως, χωρίς μια γενικότερη, ευρύτερη κοινοτική υποστήριξη, χωρίς μια κοινοτική δράση, το όλο φαινόμενο είναι πολύ δύσκολο να σταματήσει. Το πρόβλημα που το πείσαμε είναι ότι όσον αφορά τη ρύθμιση της διοκτησίας γης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εκεί αντιμετωπίσουμε πολύ μεγάλο κατακαιρματισμό όσον αφορά τις αρμοδιότητες καθώς επίσης υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά όσον αφορά το χαρακτηρισμό της γης. Αν θεωρείται αγροτική η γη, τότε την χάνει διαχείριση από την κοινή γεωργική πολιτική. Αν θεωρείται απλώς χώρος διαβίωσης, τότε αποτελεί αντικείμενο της νομοθεσίας χωροταξίας του κάθε κράτους μέλους ξεχωριστά. Θεωρήσαμε λοιπόν ότι ε, ο κατακαιρματισμός αυτός που υφίσταται αυτή τη στιγμή δεν μας επιτρέπει να έχουμε μια σφαιρική, ολιστική προσέγγιση που θα μας επέτρεπε να επιλύσουμε το πρόβλημα της υφαρπαγής γεωργικών γεών. Προτείναμε λοιπόν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενδεχομένως να κάνει μια σύσταση όσον αφορά το ζήτημα της υφαρπαγής γεών και να βασιστεί ενδεχομένως ε, στις κατευθύνσει γραμμές για την ε, υπεύθυνη έγκυο ιδιοκτησία που ήδη υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ξέρετε ότι θα μπορούσαμε κατά αυτόν τον τρόπο να διαχειριστούμε πολύ πιο υπεύθυνα την ιδιοκτησία γης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα ακόμα ερώτημα είχε να κάνει με τη δράση των ίδιων των κρατών μελών όσον αφορά αυτά τα tenure guidelines, τις κατευθυντήριες γραμμές για την έγκυο ιδιοκτησία. Ξέρετε ότι αυτές ακολουθήθηκαν πάρα πολύ κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων που είχαμε στο παρελθόν για την κοινή γεωργική πολιτική και να πρόκειται τώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση βέβαια να ελοποιήσει τις ε, κατευθυντήριες γραμμές. Ξέρετε ότι ε, ένας ε, αναλυτής μας είχε πει ότι ενδεχομένως να, υπάρχει μια μεροληπτική εφαρμογή αυτών των κατευθύνων γραμμών. Πολλές φορές επιβάλλουμε μόνο στις αναπτυσσόμενες χώρες, ενώ δεν εφαρμόζονται τόσο πιστά στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν γνωρίζω ακριβώς πώς εφαρμόζονται αυτές οι κατευθύνες γραμμές στην Ευρώπη. Ξέρω ότι η Γερμανία και οι κάτω χώρες έχουν αναλάβει κάποιες πρωτοβουλίες και προσπαθούν να δουν πώ θα καταφέρουν να χρησιμοποιήσουν επιτόπου αυτέ τι κατηβίδε γραμμέ η κάθε χώρα ξεχωριστά. Ενδεχομένω θα μπορούσαν να πνευστούν και άλλα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση από αυτό το θετικό παράδειγμα. Όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα τώρα και τη χρονική διάρκεια αυτών των συμβάσεων εξαγορά γη, Κοιτάξτε, ω προ αυτό εμεί δεν κάναμε κάποια χρονική σύγκριση αναέτο αυτών των συμβάσεων εξαγορά γη. Πάντω από ό,τι φαίνεται, Αυτές οι συμβάσεις αγοράς γης μεγάλης κλίμακας έχουν σίγουρα αυξηθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν δείτε την σελίδα 21 στη μελέτη μας, εκεί πέρα θα δείτε έναν πίνακα, μια γραφική παράσταση, την οποία έχουμε πάρει από την έρευνα Factors Markets, όπου φαίνεται η όλη αυτή τάση μεταξύ του 2003 και του 2008 όσον αφορά αυτές τις συμβάσεις εξαγοράς γης μεγάλης κλίμακας. Βλέπουμε επίσης ότι υπάρχουν κάποιες πληθωριστικές πιέσεις που έχουν αυξήσει την τιμή της γης, ιδίως από το 2007 και το 2008 και μετά, όπου οι τιμές αυτές επηρεάστηκαν και από τη γενικότερη κρίση στις τιμές των γεωργικών προϊόντων, οι οποίες είχαν εκτιναχθεί την περίοδο εκείνη. Όσον αφορά τώρα την κατανομή των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, όταν λέμε δηλαδή ότι υπάρχει πολύ μεγάλη συγκέντρωση τέτοιων γεωργικών εκμεταλλεύσεων και βλέπετε εδώ πέρα μια κατανομή και κάποια αριθμητικά δεδομένα. Πάλι στη σελίδα 24 της μελέτης μας βλέπετε ότι σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat ο ορισμός των μεγάλων γεωργικών εκμεταλλεύσεων που είναι αυτές δηλαδή που είναι από 100 εκτάρια και πάνω αντιστοιχούν στο 0,6% του συνόλου των γεωρικών εκμεταλλεύσεων, αλλά αντιστοιχούν στο 1,5 τη κερδοφορία και τη παραγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι μολονότι ο αριθμό μπορεί να είναι μικρό, η επιρροή που έχουν είναι πολύ μεγάλη. Ολοκληρώνω στο σημείο αυτό, πιέζει άλλωστε και ο χρόνο. Να προσθέσω κι εγώ κάποια στοιχεία. Όντω ακούσαμε διάφορα ερωτήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τα δεδομένα που χρησιμοποίησαμε από τα κράτη-μέλη και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλησαμε επίση να δούμε ποιο είναι ο ορισμό του ενεργού καλλιεργητή. Στα πλαίσια τη κοινή γεωργική πολιτική, τα κράτη-μέλη αποφασίζουν γι' αυτό και αυτό έχει οδηγήσει όμω σε πολλά προβλήματα. Ξέρω ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο υπάρχουν αντιδράσεις, για παράδειγμα από την Ρουμανία. Δεν καταφέραμε όμως εμείς να δούμε ακριβώς ποια είναι η πολιτική που ακολουθεί η Ρουμανία και ποια είναι η μονομένη πολιτική που ακολουθούν άλλα κράτη-μέλη όσον αφορά αυτόν τον ορισμό του ενεργού καλλιεργητή. Επικεντρωθήκαμε περισσότερο σε κάποια σωρευτικά ευρωπαϊκά δεδομένα και θελήσαμε να χρησιμοποιήσουμε δεδομένα τα οποία θα μπορούσαν να ήταν άμεσα συγκρίσιμα μεταξύ κρατών μελών. Σε ορισμένα κράτη-μέλη μπορούμε να ομαδοποιήσουμε τα στοιχεία, αλλά πάλι όχι. Πάντω επικεντρωθήκαμε περισσότερο στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο ορισμό πάντω του ενεργού καλλιεργητή, του ενεργού γεωργού, αποτελεί σημαντικό διακύβευμα τη κοινή γεωργική πολιτική. Επίση, να αναφερθώ και στι χώρε Ανατολική Ευρώπη. Είναι σαφέ ότι το 2004 όταν προσχώρησαν οι χώρε αυτέ στην Ευρωπαϊκή Ένωση είχαν μια γεωργική διάρθρωση η οποία ήταν κάπω χαοτική. Θα έλεγα λοιπόν ότι ε, η έκθεσή μας προσπαθεί να εντοπίσει κάποιους ε, πολιτικούς στόχους προκειμένου αρμονικά να διαρθρωθούν εκ νέου αυτές οι γεωργικές πολιτικές μονομένες των κρατών μελών, θα μπορούσαμε να βασιστούμε περισσότερο στην πολιτική που έχει ακολουθήσει η ΦΑΟ όσον αφορά την διάρθρωση της γεωργικής γης. Όσον αφορά τώρα την ε, άμεση κατανομή των άμεσων γεωργικών ενισχύσεων, προφανώς υπάρχουν πολύ μεγάλες ανισότητες και εμείς αυτό το οποίο προτείνουμε μέσω της μελέτης μας είναι να επανεξισορροπήσουμε την κατανομή των γεωργικών αυτών ενισχύσεων. Σε καμία περίπτωση θέλουμε να καταργήσουμε τις μεγάλες γεωργικές εκμεταλλεύσεις, ανταυτού θέλουμε να βοηθήσουμε τις μικρές εκμεταλλεύσεις που έχουν περισσότερη ανάγκη από ενίσχυση. Πολλά ερωτήματα ακούστηκαν, δεν μπορώ να τα καλύψω όλα, επομένως ολοκληρώνω σε αυτές, με αυτές τις γενικές παρατηρήσεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Νομίζω την κρίμα που δεν ακούσαμε απαντήσεις ε, σε όλα τα ζητήματα, αλλά ήταν τόσο εμπεριστατωμένη η αρχική παρουσίαση που νομίζω ότι έχουμε θίξει όλα τα ζητήματα. Μπορούμε να συναγάγουμε κάποια συμπεράσματα, θα εμβαθύνουμε σε κάποια ζητήματα, θα μπορέσουμε να απαντήσουμε τις ανάγκες που υπάρχουν για άλλες εκθέσεις ή άλλα μέσα. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας εδώ. Νομίζω ότι το θέμα αυτό όμως ε, χρήζει περαιτέρω και σε βάθος ανάλυσης μεταξύ άλλων και των πηγών. Γιατί εντάξει, κάποιες φορές μπορεί να υπάρξει μια πανεπιστημιακή μελέτη και μετά κάποια στιγμή ε, κάποιο παραπέμπει σε αυτήν και αρχίζει να έχει μια ανεξάρτητη αυτοτελή ζωή ξαφνικά. Αλλά δεν αντικατορίζει απαραίτητα και την ε, πραγματικότητα ενδεχομένω. Σα ευχαριστούμε πολύ για τα πολύ ενδιαφέροντα που μα είπατε και σίγουρα θα επανέλθουμε. Α περάσουμε τώρα στο σημείο 12. Έκθεση ζωοτεχνικών και γενολογικών όρων. Να δώσουμε απευθεία τον, ρόλο, τον λόγο συγγνώμη, στον εισηγητή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, το κείμενο το οποίο εξετάζουμε ήταν για μας μια καλή ευκαιρία ε, να αναφέρουμε τον ε, ρόλο των ζώων αναπαραγωγής. Αυτά τα ζώα σαφώς και συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη ε, περιοχών και αποτελούν βασικό πυλώνα της επιστημικής ασφάλειας στην Ευρώπη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλησε να ομοδοποιήσει όλες τις ε, οδηγίες που αφορούν ε, τους ζωοτεχνικούς όρους σε ένα μόνο νομικό σώμα υπό τη μορφή αυτού του κανονισμού. Όμως δεν διευκρινίζει τα πράγματα στο το κείμενο, σε αντίθεση με τα όσα νομίζαμε στην αρχή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει μια νέα, πιο αναρμανισμένη διάρθρωση ε, των ε, ζώων αυτών σε συγκεκριμένα είδη, το οποίο θα έχει σημαντικό αντίκτυπο για τους ακτινοτρόφους και περαιτέρω ε, οικονομικούς φορείς. κάποια στοιχεία θα πρέπει να διευκρινιστούν, μη σας πω, και αναθεωρηθούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αρχικά, θα ήθελα ε, να προσθέσουμε κάποιους ορισμούς, ιδίως σε ό,τι αφορά το είδος ε, race, ε, το οποίο δεν ορίζεται πιο συγκεκριμένα στο σχέδιο κανονισμού. Μετά, η ανταγωνιστικότητα. Οι αύξηση της ανταγωνιστικότητας θα μπορούσαν να αυξήσουν τις εξαγωγές αυτών των ειδών και αυτό το κείμενο θα μπορούσε να διευκολύνει αυτή τη διαδικασία. Ωστόσο, αυτή η φιλοδοξία δεν πρέπει να θέτει σε κίνδυνο τα μικρά σπάνια είδη ε, πολύ χαμηλού πληθυσμού ε, που αποτελούν πολύ σημαντικό τμήμα τη βιοπικιλότητα στην Ευρώπη. Θα πρέπει να διατηρηθεί αυτή η ισορροπία σε ολόκληρο το κείμενο και θα ήθελε οι αρμόδιε αρχέ να έχουν τη δυνατότητα να αρνηθούν αυτό το, την εισαγωγή ενό οργανισμού επιλογή, εάν θεωρούν ότι διακυβεύεται η γενετική βιοπικιλότητα σε μία περιοχή. Τέλο κάτι το οποίο μου είναι ιδιαίτερα προσφυλές, αλλά δεν το ε, έχει εξετάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ε, τι συμβαίνει σε αλληλοσυνερακή κλίμακα. Συμβαίνει πολύ λίγο σε αυτή, αυτή τη στιγμή, όμω ήδη υπάρχουν κάποιε μορφέ συνεργασία. Νομίζω ότι θα έπρεπε η Ευρωπαϊκή Ένωση να διευκολύνει τέτοιου είδου πρωτοβουλίε. Το βασικό βέβαια είναι η αξιοπιστία των δεδομένων και η διαλειτουργικότητά του. Ούτω ώστε οι επιμέρους αρχές ε, να ε, μπορούν να συνεργαστούν ε, σωστά. Δεν υπάρχει λόγος να προτείνω τώρα νέες νομοθετικές διατάξεις από αυτού, όμως θα ήθελα να πιστεύω την προσοχή σας σε αυτό το θέμα. Τέλος, ό,τι αφορά την κλωνοποίηση και την ευμερία των ζώων δεν χρειάζεται να επισημάνω τη σημασία του στήματο, αλλά κατά πόσο είναι σκόπιμο να τα εισαγάγουμε αυτά τα στοιχεία σε ένα τόσο τεχνικό και λεπτομερές κείμενο, νομίζω ότι δεν αρμόζει εδώ. Υπάρχουν και άλλα κείμενα ε, όπου θα μπορούσαμε να τα αναφέρουμε όλα αυτά. Δεν χρειάζεται να εισαγάγουμε τέτοιε διατάξει σε, αυτό το κείμενο, σε ό,τι αφορά τη σαφήνεια και κατανόηση ε, του ε, κειμένου. Εμείς ως πολίτες σίγουρα ε, θα θεωρήσουμε πολύ πιο επανάγνωστο έτσι αυτό το κείμενο. Κλείνοντα, θα ήθελα να στηρίξω τι γενικέ αρχέ ε, ε τη πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όμω από, εκεί και πέρα, σε πρακτικό και οικονομικό ε, επίπεδο, πρέπει τα πράγματα να αντικατοπτρίζονται σωστά. Υπάρχουν ιδιαιτερότητε του κάθε κλάδου. Θέλουμε να ενισχύσουμε την ευρωπαϊκή εκτενοτροφία, αλλά και να διατηρήσουμε, να διαφυλάξουμε τις μικρές, τα, τα μικρά είδη χαμηλού πληθυσμού. Ε, που αποτελούν ε, ιδιαιτερότητες σε κάποιες επικράτειες. Είναι λόγο το κείμενο, όμως υπάρχουν ιδιαιτερότητες για ε, κάποια είδη, όπως είναι για παράδειγμα η περίπτωση των υποειδών, που δεν πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε με τον ίδιο τρόπο με τα υπόλοιπα είδη σε ό,τι αφορά το γενολογικό τους δέντρο. Οι μεγάλες τα μεγάλα πιο σημαντικά είδη αλόγων γενικά ε, ε, ε, αντιμετωπίζονται σε παγκόσμιο επίπεδο από κοινού. Εμείς είμαστε ε, η έδρα αυτών των παγκοσμίων οργανισμών. Πρέπει να λάβουμε υπόψη όλα αυτά τα στοιχεία. Πρέπει να διαφυλάξουμε την βιοπικιλότητα και την ποιότητα των γενολογικών τους εγχειριδίων. Ευχαριστώ τους και όδης για την ενδιαφέρουσα συνεργασία. Ευχαριστώ και όσους με βοήθησαν για την εκπόνηση της έκθεσής μου. 25 Ιουνίου είναι η προθεσμία κατάθεση τροπολογιών. Θέλω ε, να κάνω τις συμβαστικές τροπολογίες πριν φύγω για διακοπές, γιατί μέσα Σεπτεμβρίου θα περάσουμε στην ψηφοφορία. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ. Ο κύριο Χάιτεμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Ο κύριος Χάιτεμα. Ε, ευχαριστώ για τον κύριο Ταντέν. Δυστυχώ ε, δεν μπορεί να παρευρεθεί ο συνάδελφο από την ομάδα που είναι ο αρμόδιο. Ε, θα μιλήσω εξ ονόματό του, αλλά συμφωνώ και απόλυτα με όσα λέω. Νομίζω λοιπόν ότι η σε έκανε εξαιρετική δουλειά. Θα θέλαμε να διευκρινίσουμε ότι συμφωνούμε με πολλά από αυτά που αναφέρει. Κάποιε παρατηρήσει θα θέλαμε να κάνουμε. Δεν είναι τόσο σημαντικέ, μάλλον ίσω σημασία, αλλά να τι διευκρινίσω παρόλα αυτά για να γίνει μια σωστή συζήτηση. Όπω ανέφερε ο εισηγητή, ε, ο τομέα των υποειδών δεν θα πρέπει να συμπεριληφθεί στην ίδια ανατομεθυσία. Θα πρέπει να δείξουμε προσοχή και θα πρέπει να δείξουμε προσοχή και σε άλλα είδη, στα βοηδή, στους χείρους, γιατί δεν πρόκειται για ζωά παραγωγής και έτσι λοιπόν η εκτροφή οργανώνεται με διαφορετικό τρόπο. Το έχει λάβει αυτό υπόψη ασφαλώ ο εισηγητή, αλλά ενδεχομένω να καταθέσουμε κάποιε τροπολογίε για να διευκρινίσουμε λίγο την κατάσταση. Το επόμενο στοιχείο. Για τη λειτουργία τη ενιαία αγορά. Σύμφωνο απόλυτα με τον εισηγητή. Υπάρχουν κάποιοι παράγραφοι και θα καταθέσουμε κάποιες ε, τροπολογίες για να υποστηρίξουμε τις, ε, τα είδη χαμηλού πληθυσμού για να προστατεύσουμε και την βιοπικιλότητα. Αλλά αυτό δεν θα πρέπει να αποτρέψει την αγωνιστικότητα. Θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα εισαγωγή υλικού αναπαραγωγή από άλλα κράτη-μέλη. Να μην χρησιμοποιείται αυτό δηλαδή ω δικαιολογία για να υπάρχουν εθνικά σύνορα στι ε, διαδικασίε αναπαραγωγή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτά ήταν όλα. Ευχαριστώ ο κύριο Ζεμπέγκα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ναι, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη να το γεγονό ότι η έκθεση αυτή ξεκινάει από τον απότερο στόχο μείωση της γραφειοκρατίας. Ωστόσο, υπάρχουν διάφοροι παράγοντες που άπτονται της εκτροφής των ζώων και της εμπορίας ζώων εκτροφής. Να ευχαριστήσω καταρχάς τον εισηγητή για το σχέδιο έκθεση. Συμφωνούμε με όλες τις τροπολογίες και με όλες τις ιδέες που ανέφερε ο εισηγητής. Ωστόσο, προκειμένου να αποφύγουμε τις πράξεις καταξιουσιοδότηση, θα πρέπει να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί. Αντιμετωπίζουμε κάποιες καταστάσεις όπου τα πράγματα πηγαίνουν καλά και το να αφαιρέσουμε 100% της πράξης κατά εξουσιοδότηση μπορεί να οδηγήσει σε καθυστέρηση στο μέλλον, σε ό,τι αφορά τον όρο breed, αναπαραγωγή. Προτείναμε ένα πολύ λεπτομερή ορισμό προς τον εισηγητή, αλλά τελικά συμφωνήσαμε επί του ορισμού που είχε προτείνει ο εισηγητής. Και αυτό για λογικούς, για νομικούς λόγους, γιατί όλοι ξέρουμε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να συμφωνήσουμε σε ένα καινούργιο ορισμό, είναι περίπλοκη διαδικασία και κατά δεύτερον επειδή χρειαζόμαστε μια σαφήνεια σε ευρωπαϊκό επίπεδο σε σχέση με τον όρο αυτό. Και ενδεχομένως ε, κάποια κοπάδια να βρεθούν σε μειονεκτική θέση αν αλλάξει ο ορισμός ακόμα και η, ο, η ΦΑΟ το αναγνώρισε αυτό γιατί είναι δύσκολος ο ορισμός του breed σε ό,τι αφορά τώρα το θέμα του μητρώου, της καταχώρησης. Αυτό το μητρό, όπως όλα τα μητρό, καλύπτεται από ένα γενικό σώμα για θέματα αναπαραγωγής. Αλλά υπάρχουν ε, στην ε, Ρουμανία ένα σύστημα, όπως και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου το μητρό αυτό είναι υπό τον έλεγχο της κυβέρνησης. Στο άρθρο 14 βλέπουμε ότι κάποια κράτη-μέλη έχουν ήδη μηχανισμούς επίλυσης των διαφορών. Προβλέπονται τέτοια συστήματα στην νομοθεσία τους. Εμείς συμφωνήσαμε να επεξεργαστούμε το θέμα των υποειδών σε ξεχωριστό κεφάλαιο, αλλά πιστεύω ότι είναι σημαντικό να διαλευκαθούν και τεχνικοί όροι, γιατί σε διάφορα κρατημέλη είναι διαφορετικές ε, οι ερμηνείε του όρου. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει σαφήνεια. Ευχαριστώ και τον εισηγητή και του συναδέλφου που βοήθησαν πολύ στι εργασίε μα και ελπίζουμε το συντομότερο δυνατόν να ολοκληρωθεί το έργο αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριο Χόισλινγκ, λέει ο πρόεδρο. Θα είμαι σύντομο. Να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την εξαιρετική δουλειά. Να συμφωνήσω και με αυτό που υπόθηκε ότι το θέμα είναι να μην καταλήξουμε σε μία εκτροφή που θα αποτρέψει την ποικιλομορφία στην Ευρώπη. Όχι, να την ενισχύσουμε θέλουμε την ποικιλομορφία και αυτό θεωρώ ότι είναι το πρόβλημα σήμερα. Θα πρέπει κάπου να το διευκρινίσουμε και αυτό, ότι δεν έχουμε οποιοδήποτε πρόβλημα με την τυποποίηση, την ενοποίηση. Όχι, αυτό που μας προβληματίζει είναι το να εξαφανιστούν κάποια είδη στην Ευρώπη. Θα πρέπει να υπάρχει ποικιλία. Έτσι λοιπόν συμφωνούμε απόλυτα επί της αρχής αυτής. Συμμεριζόμαστε επίσης το θέμα της ε, υγείας των ζώων, ότι θα πρέπει να τονιστεί πιο έντονα σε θέματα αναπαραγωγής. Γιατί δυστυχώς επικεντρωνόμαστε πιο πολύ σε θέματα υψηλή και της βέλτιστης ε, απόδοσης. Αλλά πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να υπογραμμίσουμε και την πτυχή της υγείας των ζώων. Ε, συμφωνούμε επίσης και με την τροπολογία υπερθμών 8 για την βιολογική ποικιλομορφία. Κατά συνέπεια θεωρώ ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε απόλυτα με τον εισηγητή στη φάση των τελικών διαβουλεύσεων. Είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Merci, Ευχαριστούμε κύριο Σάγνιου. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εδώ πέρα αναφερόμαστε σε ένα νέο κανονισμό όσον αφορά τις ενώσεις εκτροφέων που μπορεί να πειράσουν πάρα πολύ τα δεδομένα στον Ηνωμένο Βασίλειο, την χώρα μου. Νομίζω ότι υπάρχει μια κάποια σύγχυση ως προς το αν ο κανονισμός αυτός επιτρέπει την εξωτερική ανάθεση των προγραμμάτων αναπαραγωγής από αυτές τις ενός εκτροφέων, ορισμένες ενός εκτροφέων θεωρούν ότι θα περιοριστούν από τον κανονισμό αυτόν, άλλες πάλι όχι. Θα ήθελα μια διευκρίνηση λοιπόν ως προς αυτό. Και το πιο σημαντικό, υπάρχει αρκετό πεδίο εφαρμογή στον κανονισμό αυτό, προκειμένου οι εκτροφεί αυτοί να ακολουθήσουν ένα πρόγραμμα αναπαραγωγή, το οποίο ενδεχομένω να αντιτίθεται στο πρόγραμμα παραγωγή των επίσημων ενώσεων εκτροφέων. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Για παράδειγμα, θα πρέπει επίσημα να αποτελούν ένωση εκτροφέων προκειμένου να ακολουθήσουν ένα πρόγραμμα αναπαραγωγής. Να σας δώσω ένα παράδειγμα από τη χώρα μου έχουμε ένα, μια ένωση εκτροφέων από το Yorkshire του Ηνωμένου Βασιλείου που προσπαθούν να διασταυρώσουν βρετανικά ζώα με αμερικανικά ζώα. Σύμφωνα με τον κανονισμό αυτόν δεν θα επιτρεπόταν κάτι τέτοιο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει λάβει υπόψη τις τέτοιες περιπτώσεις. Ευχαριστούμε. Ο κ. Βαγκόντεν από την Γενική Διεύθυνση Υγείας Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για την τελευταία έκθεση που καταδεικνύει με σαφήνεια πόσο ενδιαφέρεται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το θέμα αυτό και όχι μόνο σε ό,τι αφορά τους γενετικούς ε, πόρους, ε, τα είδη και τη γενετική ποικιλομορφία, αλλά και προκειμένου να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον που να ενθαρρύνει γενικά την ε, αναπαραγωγή στην Ευρώπη. 156 τροπολογίες έχει με, λοιπόν λάβει. Να ευχαριστήσω καταρχάς τον κύριο Νταντάμ για τις ε, πολλές προτάσεις που κατέθεσε και τις πολλές τροπολογίες που θα μπορούσε να αποδεχθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να διευκρινιστεί το κείμενο και να βελτιωθεί η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ωστόσο υπάρχουν κάποια θέματα τα οποία στην παρούσα φάση θα πρέπει να τα εξετάσουμε πιο ενδελεχώς στους κόλπους της υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πέντε αναφέρω. Η εισαγωγή εκ νέου της δυνατότητας ε, απόρριψης ε, του αιτήματο αναγνώρισης ε, επιπρόσθετων εταιριών ε, αναπαραγωγής ε, κατά δεύτερον η αφαίρεση της δυνατότητας ε, για πράξη κατεξουσιοδότησης για ζώα αναπαραγωγής άλλων ειδών. Τρίτον, η αφαίρεση μεγάλων δυνατοτήτων έγκρισης πράξεων κατεξουσιοδότησης για να προσαρμοστούν τα υφιστάμενα τεχνικά προσαρτήματα κατά τέταρτον, ο περιορισμός των αποδοτικών ελέγχων πέμπτον και τελευταίο, η αποκλειστική εφαρμογή εθνικού δικαίου για την επίλυση ε, διενέξεων. Το πιο σημαντικό για την ομαστική διαδικασία είναι η στενή συνεργασία που χρειάζεται μεταξύ των θεσμικών οργάνων. Τονίζω και επαναλαμβάνω ότι οι υπηρεσίε μα στο παρελθόν και στο μέλλον θα συνεχίσουν να είναι στη διάθεση του Κοινοβουλίου για να βοηθήσουν ε, όπου αυτό είναι απαραίτητο και δυνατό για να καταλήξουμε σε ένα πολύ ισορροπημένο κείμενο με τη συνεργασία του συνομοθέτη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εμείς σας ευχαριστούμε. Ο κύριος Νταντάν τώρα να πάρει το λόγο για να κλείσουμε και τη συζήτηση αυτή. Ναι, ευχαριστώ Πρόεδρε. Καταρχάς να ευχαριστήσω όλους τους εκπροσώπους των πολιτικών ομάδων για τα σχόλια τους. Όντως, Νομίζω ότι θα μπορούσαμε να καταλήξουμε σε μια συμφωνία. Έχουν αρχίσει να συγκλίνουν πολλοί απόψεις μας. Απλώς ε, να διαβεβαιώσω τον συνάδελφο Άγνιου ότι προφανώς η Ευρώπη λαμβάνει υπόψη της την διαφορετικότητα που υπάρχει επιτόπου σε κάθε κράτος μέλος. Άρα στο παράδειγμα το οποίο έθεσε δεν υπάρχει κανένα εμπόδιο στο κείμενο προκειμένου να γίνει αυτό το οποίο περιέγραψε. Άκουσε επίση και τι παρατηρήσει Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, Ω ε, εισηγητή και στην Επιτροπή Περιβάλλοντος ε, έχω συνεργαστεί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έχουμε καταλήξει σε συμφωνίε. Νομίζω ότι το ίδιο συνενετικό πνεύμα θα πρέπει να έχουμε και εδώ πέρα με την έκθεση αυτή στην Επιτροπή μα. Είπα πριν από λίγο ότι το Συμβούλιο προχωρά και αυτό παράλληλα με εμά και ότι ήδη εκ μέρους του Συμβουλίου έχουμε κάποιες προτινόμενες διατυπώσεις που θα μπορούσαν ήδη να διευκολύνουν την εργασία που προτιθέμεθα να κάνουμε στα πλαίσια του τριμερούς διαλόγου. Όσον αφορά πιο συγκεκριμένα τις κατεξοδότηση πράξης, ξέρετε ότι αρχικά το κείμενο προέβλεπε ένα πολύ μεγάλο αριθμό τέτοιων πράξεων. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ήδη μία σημαντική εμπειρία στον τομέα αυτό των ε, κατεξόντων πράξεων και θεωρήσαμε ότι το βασικό κείμενο θα πρέπει να είναι αρκετά σαφές ώστε να λειτουργήσει απλώς και μόνο με εκτελεστικές πράξεις. Υπάρχει και ένα ευαίσθητο βέβαια ζήτημα, το ζήτημα της διεύρυνσης σε άλλα είδη. Το κείμενο το οποίο σας παρουσιάστηκε έχει να κάνει με τα βοηδή, τα χειροειδή, τα εγωπρόβατα. Ξέρετε ότι υπάρχουν όμως και πολλά άλλα είδη. Και κυρίως τα πουλερικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρούσε ότι θα μπορούσε να καλύψει και όλα αυτά τα είδη μέσω κατεξότηση πράξεων. Το Συμβούλιο ζήτησε νομοθετική πράξη για τα υπόλοιπα είδη που δεν καλύπτονται από αυτόν τον κανονισμό. Νομίζω ότι και εμείς ακριβώς αυτό θα πρέπει να ζητήσουμε, συγκεκριμένη ξεχωριστή νομοθετική πράξη για τα υπόλοιπα είδη. Το ζήτημα είναι πολύ σημαντικό. Μίλησα και με τους σκιώδεις εισηγητές και δεν νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε πίσω σε αυτό το ζήτημα. Σας ευχαριστώ πολύ και εκ των προτέρων σας ευχαριστώ για τη μελλοντική συνεργασία που θα έχουμε. Κύριε Μπούντα, θέλετε κι εσείς τώρα το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όσον αφορά αυτούς τους οργανισμούς αναπαραγωγής. Νομίζω ότι θα πρέπει να επισέλθουμε σε λίγο περισσότερες λεπτομέρειες, προκειμένου να έχουμε και εμείς περισσότερες πληροφορίες από αυτούς τους οργανισμούς αναπαραγωγής, breeding bodies. Όταν μια γεωργική εκμετάλλευση εισάγει κάποια ζώα, θα πρέπει να γνωρίζει ότι τα στοιχεία τα οποία λαμβάνει από τον πολίτη όντω αντιστοιχούν στην πραγματικότητα. Ξέρετε ότι πολύ συχνά στο παρελθόν πολλέ από τι πληροφορίε που δίνει ο πολιτή δεν συνάδουν ε, με την πραγματικότητα και η ποιότητα τελικά του ζώου που αποτέλεσε αντικείμενο πόλη ήταν πολύ χαμηλή, πολύ χαμηλότερη από αυτή που λεγόταν στο δελτίο το οποίο τον συνόδευε, ο κύριο Νταντά. Ναι, μα συμφωνώ με τον κύριο Μπούντα. Τα στατιστικά δεδομένα, μάλλον οι ε, στατιστικολόγοι μιλούν για τη λεγόμενη διάρκεια βιωσιμότητα των δεδομένων. Αυτό θα πρέπει να μας απασχολήσει. Θα πρέπει δηλαδή να μπορούμε από τη μία χώρα στην άλλη να έχουμε αξιόπιστα συγκρίσιμα δεδομένα, προκειμένου να διασφαλίζεται πλήρω ο καταναλωτή, ο πελάτη. να αγοράζεται ένα ζώο θα πρέπει να σε θέσει άμεσα να ξέρετε τι χαρακτηριστικά έχει και πώς μπορεί αυτό να καταχωρηθεί στα εθνικά βιβλία αναπαραγωγής. 25 Ιουνίου στις 12 το μεσημέρι καταληκτική προθεσμή για την υποβολή τροπολογιών. Και εξ ονόματος Πρόεδρου να ζητήσω τώρα από τους συντονιστές να παραμείνουν στην αίθουσα για τη συνεδρία των συντονιστών. Σας ευχαριστώ πολύ.